Yes, hello everyone. Uh, we can... Καλό απόγευμα σε όλους. Να συνεχίσουμε. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βέλα, τον Επίτροπο Βέλλα. σχετικά με την αλίευση παρανόμων ειδών Γνωρίζετε ότι έχουμε δεσμευθεί μάλλον το κυνήγι παρανόμων ειδών, έχουμε δεσμευθεί σε, μια, σε ένα συνολικό πλαίσιο προστασίας όλων των ειδών πτηνών. Είχαμε και την οδηγία Habitat για την προστασία της βιοπικιλότητας και όλων των μεγαλόσωμων σαρκοβόρων ειδών, όπως και των οικοσυστημάτων τους. Πρόκειται για θέμα πολύ επίκαιρο σε πολλές χώρες. Στη Ρουμανία έχουμε μεγάλους πληθυσμούς μεγάλων σαρκοβόνων συμπεριλαμβανομένων ειδών αρκούδας. Το 35% συνολικά των λύκων στην Ευρώπη και ένα σημαντικό ποσοστό λίγκα σαρκοβόρα είδη που πολύ συχνά έρχονται σε επαφή με τις περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι σημαντικό επομένως να έχουμε, να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της συνύπαρξής μας με μεγάλες σαρκοβόρα είδη. Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε τον Επίτροπο που βρήκε το χρόνο να έρθει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα που είναι σημαντικό για τους πολίτες των χωρών μας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση σας δίνω το λόγο κύριε Βέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα στα μέλη. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική η παρουσία σας καθ' όλη τη διάρκεια της εντολής μου για την προστασία του οικοσυστήματός μας και ιδιαίτερα στους φακέλους αρμοδιότητάς μου. Αυτό ήταν απόλυτα προφανές στο fitness check της προστασίας ε, των οικοσυστημάτων και με το σχέδιο δράσης παρουσιάσαμε και για την οικονομία και για τους πολίτες και για το οικοσύστημα. Αποστήλατε ένα σημαντικό μήνυμα προς την Κομισιόν και επηρεάσατε τα πορίσματα του fitness check είναι σαφές ότι έχουμε μια κοινή δέσμευση για να προστατεύσουμε την ε, φυσική, το φυσικό κλειοδότημα ή ε, στην Ευρώπη και υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη να αναλάβουμε δράση προς την κατεύθυνση αυτή ε, δεδομένης της κατάστασης της βιοπικιλότητας του 60% της μείωσης που ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, έχει σημειώσει στην, στην έκθεση του 2018, όπως και την ταχύτατη μείωση των πληθυσμών σε συγκεκριμένα είδη. Όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολο να τα αποδεχθεί κανείς και σοκάρουν και είναι αρκετά εκπληκτικό ότι ακόμα και εν ώψη τόσο δυσχερών εκθέσεων διστάζουμε ακόμα να λάβουμε δράση. Όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την ε, ευζοία αλλά και την ασφάλεια την επισητιστική μας για την ίδια μας την επιβίωση. Ένα απίστευτο 70% του συνόλου των ειδών και ο άνω του 80% των οικοσυστημάτων μας βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση υγείας. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος αλλά περιορισμένη και επιμέρους μικρής κλίμακος συνολικά. Επομένως, δεν μπορεί ο πλανήτης να παραδώσει επί των στόχων που είχαν συμφωνθεί για το 2010 για την προστασία της βιοποικιλότητας. Πέρυσι στο Σαρμεσέικ, στην COP14, ε, σημειώσαμε ότι πρέπει να επιταχύνουμε την ε, δραστηριότητά μας για το πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020 που θα συμφωνηθεί του χρόνου στο Πεκίνο στην COP15. Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει πλέον μια όθηση για ένα New Deal για τη φύση. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να θυμηθούμε και τον Sir David Attenborough σχετικά με τους μηχανισμούς καταστροφής που έχουμε στήσει παντού. Είναι θετικό για παράδειγμα ότι βλέπουμε ότι η Γαλλία θέλει να κάνει την προστασία της βιοποικιλότητας κατά την προεδρία του G7 υψηλής προτεραιότητας. Άλλη μια σύνοδος βιοποικιλότητας ε, σχεδιάζεται για την Γενική Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών το 2020, για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ηγείται σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να συνεχίσει να προστατεύει και να ε, αυξήσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οικοσυστημάτων. Είναι το μοναδικό απαραίτητο και άρτιο νομικό πλώσιο για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Δεν χρειάζομαι μόνο την προστασία των περιοχών Natura 2000, αλλά πολύ περισσότερο στην προσπάθεια των επιπολιαστών, στην ε, προσπάθεια της ενσωμάτωσης των ε, της λήψης μάλλον υπόψη των οικοσυστημάτων στην ε, διαδικασία διαμόρφωση πολιτικής και λήψη απόφασης. Και σε ανταπόκριση προς τα πορίσματα του fitness check θα πρέπει να εστιαστούμε στα θέματα υλοποίησης, ιδιαίτερα μέσω του σχεδίου δράσεως για την φύση, τους πολίτες και την οικονομία. Πολλές από τις σχεδιαζόμενες δράσεις ήδη έχουν εγκατασταθεί και είμαι, έχω εμπιστοσύνη ότι το σχέδιο δράσης αυτό θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η δέσμευση από πλευρά σα υπήρξε εξαιρετικά χρήση μέχρι εδώ. Πολλέ από τι προκλήσει αυτέ πρέπει να αντιμετωπιστούν τοπικά και περιφερειακά μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών διευκολύνεται σημαντικέ δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί στο εδαφο η πρώτη επιτυχία που θέλω να σημειώσω είναι η αύξηση του, ε, της χρηματοδότησης κύκλου ζωής ε, κατά 10% και για την προστασία των ειδών. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη επικαιροποίησει τα πλαίσια δράσης τους και συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων επένδυσης για είδη ζώων και οικοσυστήματα για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Επίσης, έχουμε την οδό της ε, επιβολής και επικύρωσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές Natura 2000. Πολλά κρατημέλη έχουν μείνει πίσω στην περιοχή αυτή, αλλά οι προσπάθειές μας νομίζω ότι αρχίζουν και καρποφορούν με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών αυτών να, έχουν, να ανέρχονται πλέον στο 70%. Ήθελα επίσης να αναφερθώ στα θέματα της συζήτησης και του διαλόγου. Η Κομισιόν έχει σχεδιάσει και συνεχίζει διμερείς επαφές με ενδιαφερόμενους φορείς και κράτη-μέλη, το οποίο έχει οδηγήσει σε περαιτέρω φύλλα πορείας οδικούς χάρτες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης προστασίας ο πρώτος γύρος διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς και κράτη-μέλη επί τη βάση ενός εγγράφου κατευθύνσεων έχει ξεκινήσει. Ο δεύτερος γύρος θα ακολουθήσει σύντομα. Το έγγραφο αυτό κατευθύνσεων θα περιλαμβάνει και παραδείγματα βελτίστων πρακτικών ώστε να διαμορφώσουν την γνώση μας και λύσεις. Προκειμένου να διευκρινίσουμε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ιδιαίτερα την ευελιξία που μπορεί να περιέχει Θα παρακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση την ομολογία απολύτως πιστά του δικαστηρίου. Ωστόσο υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας και είναι η πρόθεσή μας να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, τη γνώση, την ενημέρωση σχετικά με τα περιθώρια αυτά ευελιξίας που υπάρχουν. Σε Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Φιλανδία, Γερμανία και Γαλλία έχουμε προσχεδιάσει διάφορες εκδηλώσεις και διάφορες επαφές γιατί ο καλύτερος τρόπος να μειώσουμε τις ε, αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις είναι να συζητούμε μεταξύ μας. Τον μήνα αυτό είχα την ε, ευκαιρία να απευθυνθώ και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ε, το σχέδιο δράσης για τους πολίτες και την οικονομία προβλέπει μέτρα για την προστασία των ε, σαρκοβόρων ειδών μεταξύ άλλων και μετά την έγκριση του σχεδίου αυτού δράσεως εγώ κατεύθυνα τις υπηρεσίες μας ε, να διοργανώσουν ad hoc συναντήσεις επιτόπου αποδεχόμενοι προσκλήσεις από τοπικές και περιφερειακές ε, διοικήσεις από την Επίτροπο των Περιφερειών ώστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σχετικά με την προστασία συγκεκριμένων ειδών από συγκεκριμένες περιφέρειες Ισπανίας, Γερμανίας, Ρουμανίας, εξετάζοντας, αναζητώντας πρακτικές λύσεις δυσκολίας ελοποίησης εντός του παράντος πλαισίου. Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι και επομένως με χαρά βλέπουμε την ε, αξιολόγηση ομοτήμων που σχηματίζεται σιγά σιγά. Εδώ το σκεπτικό είναι να αυξήσουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μιλών και μεταξύ διαφόρων επιπέδων αρχών σε διάφορα κράτη που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Για παράδειγμα, η Ισπανία χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό και επισκεπτόμενοι την Γαλλία για να ανταλλάξουν ε, ε, ε, ενημέρωση για το σχέδιο διαχείρισης της προστασίας του γαλλικού λύκου είναι ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Καλύπτουμε συνολικά άνω των 1.500 ειδών και μόνο λίγα από αυτά αποδεικνύονται ιδιαίτερα προβληματικά για τη συνύπαρξη με τους ανθρώπους. Τα μεγαλόσωμα σαρκοβόρα πράγματι εγείρουν ανησυχίες σε κάποιες από τις περιφερειές σας, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την κατεύθυνση του λόγου για τον οποίο χρειάζονται προστασία. Οι λύγκες, οι λύκοι, οι αρκούδες είναι απόλυτο αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής μας, του οικοσυστήματος, της παράδοσης της βιοπικιλότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή και που αντιμετωπίζει η ε, υπαρξιακή απειλή. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα που σας ανέφερα και περισσότερα, αλλά τελικώς από τις τοπικές και κρατικές αρχές θα εξαρτηθεί να καλύψουν τις ε, περιφερειακές και τοπικές ανάγκες. Τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης ή ανάκτησης αναλόγως προς το καθεστώς, την κατάσταση του αποθέματος του κάθε είδους. Αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις και να εφηγραμμίζονται και με την ευρωπαϊκή αλλά και με τις εθνικές νομοθεσίες. Αυτό ήταν το μήνυμα που απέστειλα με τον Επίτροπο Χόγκαν στους ε, Υπουργούς ε, Γεωργίας και Περιβάλλοντος στην κοινή μας συνάντηση της 11 Φεβρουαρίου και ελπίζω να υποστηρίζετε τη θέση μας. Και να σας πω λίγα λόγια για τα πουλιά. Σχέδια δράσης έχουν αναπτυχθεί για 16 είδη πουλών συμπεριλαμβανομένου λαμβανομένης της 18 Έχουμε διάφορα είδη που απειλούνται και οι υπουργοί καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης με μορατόριου ε, μορατόριουμ της εποχής κυνηγιού και η Κομισιόν επικαιροποιεί επίσης ένα έγγραφο βασικών σκεπτικών για την περίοδο αναπαραγωγής και μετανάστευσης των ειδών που των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μια πιο συνεπή προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζουν ότι η περίοδος κυνηγιού δεν θα τοποθετείται στην περίοδο κατά την οποία τα είδη είναι πιο ευαίσθητα. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές αιτίες της μείωσης των πληθυσμών των ειδών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι όπως προβλέπει η νομοθεσία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκίνησα λέγοντας ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προστατεύσουμε την βιοεπικλαιότητα. Θα προσθέσω τους εξή. Καταρχά, οι πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρώπης. Το πιο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του 2018 επιβεβαιώνει εκ νέου πόσο πραγματικά ανησυχούν και ενδιαφέρονται οι πολίτες για την Ευρώπη. Το 96% των απαντήσεων θεωρούν ότι έχουμε μια ευθύνη να προστατεύσουμε τη φύση. Και το 93% συμφωνούν ότι η υγεία και η ευζοία μας εξαρτάται από την φύση και την βιοποικιλότητα. Ο δεύτερος λόγος που θέλω να σας αναφέρω είναι η συνεχιζόμενη αλλαγή του κλίματος. Η βιοπικιλότητα συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Όταν το κλίμα δυσχεραίνει, λέει ο μιλητής, χάνουμε περισσότερα είδη. Επομένω, η προστασία τη βιοπικιλότητα και των ειδών, όπω και τη κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση τη δηλαδή, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να υλοποιείται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε τι προσπάθειε αντιμετώπιση τη απώλεια βιοπικιλότητά μα, αναθεωρώντα την κοινή μας γεωργική πολιτική και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εντός του οποίου η φύση ενισχύεται, η προστασία της φύσης ενισχύεται πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας σε αυτές τις περιοχές. Στην COP15 θα έχουμε ήδη μια νέα επιτροπή και θα πρέπει ήδη από τώρα να προετοιμάσουμε το έδαφος για ένα new deal για τη φύση και το οικοσύστημα στην επόμενη περίοδο. Και επ' αυτού είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να βαστούμε στην υποστήριξή σα. Ευχαριστώ για την προσοχή και είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σα καθώ και για το ενδιαφέρον σα για το θέμα αυτό. Συνάδελφοι, από δύο λεπτά ο κάθε ομιλητή, η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι μαζί μας σήμερα. Όλοι μας εδώ ασχολούμαστε με μεγάλο ενδιαφέρον με την οδηγία για το habitat και την προστασία των ειδών. Προστασία που είναι όλο και πιο απαραίτητη. Έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις και μελέτες που μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Στην δική μου τη χώρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθούμε παράδειγμα γιατί 64 είδη ε, πουλιών που απειλούνται είναι ανοιχτά στο κυνήγι. Εγώ θα ήθελα να ξέρω λοιπόν και τη δική σας άποψη από αυτού, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στα μεγαλόσωμα σαρκοβόρα και πάνω απ' όλα στον λύκο, που ως είδος προστατευμένο ε, βρίσκεται σε υπερπληθυσμό σήμερα. Σε ένα βαθμό λοιπόν προστατεύεται από την οδηγία Habitat και αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα σε κάποιες περιφέρειες των Άλπαιων. Ιδιαίτερα των Γαλλικών Άλπαιων. Η προστασία του λύκου είναι πρόβλημα για τους εκτινοτρόφους και για συγκεκριμένες ε, περιφέρειες κτηνοτροφίας που αισθάνονται την ε, πίεση της παρουσίας του λύκου στην οικονομική τους δραστηριότητα, στις οικογένειές τους, στη ζωή τους. Και παρά τα μέτρα συνοδείας, παρά την, την αδειοδότηση συγκεκριμένων περιόδων ε, θανάτωσης, ε, εν περιπτώσει μείωσης του πληθυσμού, ε, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Εγώ λοιπόν ήθελα να υπογραμμίσω το πρόβλημα του λύκου πρέπει να εξακολουθήσουμε να θεωρούμε ότι είναι προστατευόμενο είδος ή θα πρέπει να έχουμε μια διαχείριση λίγο πιο ευέλικτη για το είδος αυτό. Thank you very much. Uh, now, Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μελιόρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτρο, χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε το σημαντικό θέμα της βιοπικιλότητας. και θα συμφωνήσω με την κυρία Γκροστέτ. Έχω ερωτήσει σχετικά με τον Λίκο. διότι στο Βραντεμβούργο που είναι το δικό μου το κρατήδιο, Έχουμε πάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού του λύκου της, ε, όλης της ε, Γερμανίας και καταλαβαίνετε ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα. Η μόνιμη επιτροπή συνεδρίασε τον Νοέμβριο του 2018 στο Στρασβούργο και πρότεινε ε, να περάσει ο λύκος από ε, το παράτημα 2 στο παράτημα 3. Ε, έτσι μπορεί να αποτελέσει και θύραμα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αν θα στηρίξει αυτό το αίτημα που έχει αναβληθεί. Εάν αν όχι, γιατί. Και τώρα που μιλάμε για τον Λύκο, Χρειαζόμαστε αξιόπιστα δεδομένα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ανάγκη προστασίας του λύκου. Στην επιστολή σας ε, της 11ης Φεβρουαρίου αναφέρεστε στο διάστημα 2013 έως 2018. Λέτε ότι θα υποβληθούν τα σχετικά δεδομένα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πότε θα γίνει αυτό. Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένο μήνα του έτους διότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός. Αν ε, δηλαδή βρίσκεται σε καλή κατάσταση ο λύκος και αν μπορεί να περάσει από το παράρτημα 2 στο παράρτημα 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ τον κύριο Γκερμπράντη, τον αντικαθιστά ο κύριος Σε Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Ε, εδώ στα έγγραφά μας ε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χάρτης που δείχνει ε, πού βρίσκονται τα σημαντικά σαρκοβόρα. Και μάλιστα δύο κράτη-μέλη έχουν και τα τέσσερα σαρκοβόρα. Ως Φιλανδοί λοιπόν και νομίζω ότι και οι Σουηδοί θα το αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, πιστεύουμε ότι έχουμε ειδική ευθύνη. Όταν όμως μιλάμε και για ειδική ευθύνη, θα θέλαμε επίσης ε, να μας αντιμετωπίσετε με κατανόηση. Ο συνάδελφός μου εδώ πέρα μου λέει ότι ένας λύκος έχει περάσει από τη Γερμανία στις κάτω χώρες. Εντάξει, ε, τέλεια είναι τα πράγματα. Στον χάρτη βλέπετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ούτε λίγκα, ούτε λίκο, ούτε αρκούδα, ούτε αδιφάγους. Ε, μάλλον έχουν αρκετούς μονόκερους ε, στο θηρεό τους. Αλλά, εβάσε τόση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συχνά χώρες χωρίς εμπειρίες με σαρκοβόρα μιλούν χωρίς τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι σε μας που έχουμε το πρόβλημα. Κάτι λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι υπάρχει σαφής τάση αστικοποίησης όσον αφορά ε, τα σαρκοβόρα και στις αρκούδες και στους λύκους και στους λύγκες. Μόνο ο αδιφάγος ε, είναι πολύ ντροπαλός ε, και δεν πλησιάζει στις πόλεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζουν ε, οι συνήθειες των ζώων αυτών, μετακινούνται σε περιοχές όχι μόνο γειτονικέ σε αυτές που ζουν οι άνθρωποι, αλλά συχνά κυκλοφορούν ανάμεσα στα σπίτια στη Δυτική Φιλανδία. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση δεν υπάρχουν φυσικοί οικότοποι. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τις κάτω ε, δεν ε, είναι ούτε οι φυσικές περιοχές των κάτω χωρών ε, φυσικός οικότοπος για τους λύκους. Σας παρακαλώ να επιδείξετε κατανόηση για τα προβλήματα μας και τα μέτρα που λαμβάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ. Κατανόηση όμως ε, και απέναντι στους άλλους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριε Χόισλινγκ, δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, ας ε, μιλήσουμε λογικά για την βιοπικιλότητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε χάσει το 70% των εντόμων. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα και συνεχίζεται η τάση αυτή και συνδέεται και με τη γεωργία μας. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ε, συνομίλησα με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χόγκαν. Συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κοινή γεωργική πολιτική ε, με τον ίδιο τρόπο που φτάσαμε μέχρι εδώ. Χάνουμε πολλά μικρά πουλιά και αυτό είναι δραματικό ενώ τώρα μιλάμε για ένα είδος το οποίο ε, δυσκολεύει τη ζωή για κάποιες περιφέρειες. Νομίζω ότι είναι υπερβολική η συζήτηση σε πολλούς τομείς. Ναι, φυσικά πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον λύκο, αλλά να σας δείξω και μια άλλη στατιστική. Στη Γερμανία ε, τα πρόβατα έχουν μειωθεί κατά 50% τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό μήπως συνδέεται με τον ε, λύκο? Όχι, καθόλου. η κτηνοτροφία ε, μειώνεται διότι ε, έχουμε λάθος πολιτική προώθηση. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται υπερβολικά διότι και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μπορεί να σκοτώσει κανείς σε προβληματικούς ε, λύκους. Ε, απλά δεν είναι πολύ εύκολο να λάβει κανείς την άδεια για να σκοτώσει έναν λύκο. Ποιο είναι το πρόβλημα. το πρόβλημα είναι οι πελεκάνοι, οι ενιτρίδες. Ε, δεν μπορεί αυτή να είναι η απάντηση στα προβλήματά μας. Ε, η απάντηση θα πρέπει να είναι να έχουμε λογικά μέτρα προστασίας, ε, λογικά μέτρα αποζημίωσης και όταν υπάρχουν προβλήματα να ενεργούμε ανάλογα. Φυσικά θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε ε, μήπως αρκούν τα μέτρα μας, αλλά απέχουμε πολύ από αυτό. Η κυρία ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι περίεργο που μία συζήτηση για το κυνήγι των πουλιών στην Μάλτα έχει καταλήξει σε συζήτηση για ε, τους λύκους. Πολλά μεταναστευτικά πουλιά επιστρέφουν από την Αφρική στην Ευρώπη, τα οποία όμως ε, θα σκοτώσουν κυνηγοί, παρότι αυτό είναι παράνομο στην Ευρώπη. Και ευτυχώς η Κομισιόν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και στρέφεται κατά της ε, Φιλανδίας για το κυνήγι της πάπιας Άιντερ. Και τα ορτίκια και άλλα είδη ευάλωτα υπάρχουν πέρα από τα είδη που σκοτώνονται στην Μάλτα και μάλιστα συχνά με παράνομα εργαλεία. Για την 18 ουρα λοιπόν ε, δεν είχαμε συγκεκριμένα μέτρα, βλέπουμε όμως ότι σκοτώνονται κατά εκατοντάδες. Το... Η σεζόν του κυνηγιού ανοίγει ακριβώς τη στιγμή που ε, αρχίζουν να κυκλοφορούν 18 ε, Γιατί λοιπόν στρέφεστε κατά της Φιλανδίας και όχι κατά της δικής σας χώρας, της Μάλτας. Επίσης θα ήθελα να μιλήσω για τα μεγάλα σαρκοφάγα. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να αποδυναμωθεί η οδηγία για τους οικοτόπους και τώρα έχουμε το σύνδρομο της κοκκινοσκουφίτσας και έτσι στρεφόμαστε κατά του λύκου, του λίγκα, της αρκούδας και άλλων ειδών. Μέχρι τώρα, κύριε Επίτροπε, έχετε διατηρήσει τη γραμμή σας όσον αφορά την οδηγία αυτή. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι όλα τα φυτά και τα ζώα που εμπίπτουν στην οδηγία αυτή θα συνεχίσουν να προστατεύονται στο μέλλον συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σαρκοφάγων. Θα θέλαμε πολύ να το δούμε αυτό. Ε, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Καλό απόγευμα σε όλους. Άκουσα από διάφορους συνάδελφους, ε, εδώ είμαι, προτάσεις που βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτες. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις οδηγίες ε, γίνεται χρήση των εξαιρέσεων απολύτως απαράδεκτη στην ουσία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο επί τη βάση ε, συμφερόντων τοπικών και ιδιαίτερα φιλικών ε, προς τους κοινοτρόφους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και βλέπουμε και τις ε, καταδικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικώς. Νομίζω ότι είναι καλό νέο, καλή είδηση ότι η, η δοκιμή, το fitness check έδωσε θετικό πόρισμα για την οδηγία και επομένως δεν μπορούμε να πειράξουμε τις διατάξεις αυτές. Πρέπει να θεωρούνται απολύτως ενισχύ και κατάλληλες. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν το επίπεδο της προστασίας για τα μεγαλόσωμα σαρκοβόρα μεταξύ των οποίων τον λύκο ε, το κυνήγι ποτέ δεν είναι ε, συνεπές ε, προς την προστασία της βιοποικιλότητας. Εκεί όπου έχουμε κυνήγι, έχουμε και λαθρέο κυνήγι και επομένως δεν μπορεί κανένα σχέδιο διαχείρισης να είναι κατάλληλο. η εποχή κυνηγιού που μόλις έκλεισε στην Ιταλία είχε απολύτως αρνητικό κατάλογο γιατί είχαμε και πολλά θύματα πληθυσμού στον κόκκινο κατάλογο που προστατεύονται από τα ε, είδη, δηλαδή απαριθμούνται μεταξύ των ειδών της οδηγίας που είναι προστατευμένα και θα κλείσω με ένα μέγεθος το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τα, για τα δίκτυα ασφαλείας ε, είχαμε 84, 84 τραυματίες και 30 νεκρούς σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν και ο πρώτος κύκλος ερωτήσεων. Τώρα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο, αλλά σας παρακαλώ να ε, μην μιλήσετε πάνω από ένα λεπτό έκαστος. Ο κύριος Ντόρφμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Νωρίτερα μας κάνατε μια αρκετά περιεκτική σύνοψη, όμως δεν είδα συγκεκριμένε προτάσεις. Θα διαφωνήσω με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, ε, παρότι προέρχομαι από την ε, ίδια χώρα. Από την εποχή που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία υπήρχαν ε, περίπου 100 λύκοι στην Ευρώπη, απειλούνταν με εξαφάνιση. Τώρα ο αριθμός έχει πολλαπλασιαστεί. Νομίζω πως η οδηγία έχει επιτύχει λοιπόν το στόχο της και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και το καθεστώς προστασίας του λύκου. Επίσης, είπατε ότι όλα είναι θετικά και ότι οι εκπρόσωποι του γεωργικού κλάδου ε, αποχώρησαν από την ε, συζήτηση ακριβώς λόγω αυτής ε, της ευελιξίας. Δεν νομίζω πως έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ευελιξία έχει, δεν έχει αυξηθεί για τα κράτη-μέλη, το αντίθετο έχει μειωθεί. Να σας ρωτήσω επίσης το εξής. Ε, μας είπατε πως υπάρχουν ορισμένες περιοχές ε, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και όλα ε, βαίνουν καλώς. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες από αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πένον έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, η γρήπη των χείρων είναι η πανόλη των χείρων, ε, είναι μια τρομακτική ασθένεια για την οποία δεν υπάρχει εμβόλιο. Όμως μια μελέτη από τη Σλοβακία αναφέρει ότι εκεί όπου ζουν λύκοι υπάρχουν ελάχιστα κρούσματα πανόλης των χείρων, ενώ όπου δεν υπάρχουν λύκοι το 90, ε, παρατηρείται το 93% των κρουσμάτων. Στην Ανατολική Σλοβακία, όπου ζουν λύκοι, ε, τα κρούσματα είναι μόνο 7%. Αυτό λοιπόν ε, τι σημαίνει, ότι ο λύκος σκοτώνει τα άρρωστα αγριογούρουνα και έτσι εμποδίζει την εξάπλωση της ασθένειας. Ε, και στο Εθνικό Πάρκο του Yellowstone έχουμε δει ότι εκεί όπου επανησύχθη ο λύκος έχει αυξηθεί ε, με πολύ γρήγορους ρυθμούς η βιοπικιλότητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, η ύπαρξη του λύκου στην Ευρώπη έχει πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας συνιστούσα να το ξανασκεφτείτε πρωτού αναλάβετε οποιαδήποτε δράση. Σας ευχαριστώ πολύ που κρατήσετε το χρόνο ομιλίας. Η κυρία Σουάι και έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, τα κράτη-μέλη συζήτησαν για τα πτηνά που ζουν στην ευρασιατική ζώνη. Συζήτησαν συγκεκριμένα για την ασπρομαγουλόχυνα, ο, που είναι προστατευόμενο είδος. Ο αριθμός της όμως έχει πολλαπλασιαστεί από την ημερομηνία που ατέθησε ισχύ η οδηγία. Και χρειάζεται και η οδηγία αυτή είχε δημιουργηθεί για να προστατεύσει αυτά ε, τα πτηνά, αυτές τις χήνες. Ε, τι γίνεται όμως τώρα έχει εφαρμοστεί σωστά η οδηγία το 2019. Επίσης, θεωρείται ότι κατά την εφαρμογή του άρθρου 16 οι επιπτώσεις της ε, προστασίας του λύκου παρατηρούνται σε, όλη την, ε, σε όλες τις γύρω περιοχές. Ε, στις κάτω χώρες δεν υπάρχει χώρος για να ζήσουν λύκοι. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μέσω σχεδίων προστασίας για τον λύκο. Νομίζω πως εκεί πρέπει να εστιάσουν οι προσπαθίες μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι το οποίο ήδη ακούστηκε. Ο συνάδελφος που θεωρούσε ότι η συζήτηση αυτή αφορά μόνο τη Μάλτα. Να του πω πως όχι. Η συζήτηση αυτή αφορά το κυνήγι προστατευόμενων ειδών. Αλλά αν θέλετε να, περιοριστούμε σε μια χώρα, ας πούμε λίγο και το εξή. Εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται ανεξέλεκτα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και έλεγα στον συνάδελφο ότι είμαι μέλος της Life ε, Μάλτας και αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ε, υπάρχει περιθώριο για ανεξέλεκτες ενέργειες. Αλλά ας μην λέμε ότι για όλα αυτά η Μάλτα, ας μιλήσουμε και για την Αυστρία και για άλλες χώρες. Στη Μάλτα έχει απαγορευτεί το κυνήγι της ακαθούρας στην Άνοιξη και στο σχέδιο δράσης Βλέπουμε επίσης ότι η μείωση του πληθυσμού ορισμένων ειδών έχει να κάνει και με την ε, κατάσταση και την επιδείνωση των ε, διαιτημάτων τους, αλλά και με την γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι μέτρα έχουν γίνει για να αντιστραφεί αυτή η επιδείνωση των ε, οικοσυστημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε τώρα το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προτού απαντήσω στι συγκεκριμένε ερωτήσει, επιτρέψτε μου να κάνω μερικά γενικά σχόλια. Καταρχά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και επικρίσεις εκτό από επένου, έτσι ώστε να εστιάσουμε στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Νομίζω πως θα πρέπει να αναφερθούμε στην κρίση της βιοπικιλότητα. Διότι η απώλεια βιοπικιλότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσει που αντιμετωπίζουμε μαζί με το, την κλιματική αλλαγή. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ότι δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους για τη βιοπικιλότητα. Ωστόσο αυτό με ανησυχεί, διότι πάντα επαναλαμβάνουμε τις ίδιες δηλώσεις, έτσι πιο χαλαρά κάθε φορά, χωρίς να έχουμε πείγνωση του πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση. Εάν πράγματι θέλουμε να δείξουμε ότι ανησυχούμε, τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια. Και δεν πρέπει να το κάνουμε επιλεκτικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε με όλα τα αίτια της ε, επιδείνωσης της κατάστασης. Ξεκίνησα με μια ευρύτατη δημόσια διαβούλευση για το αν η οδηγία είναι πλέον κατάλληλη ή όχι και όπως γνωρίζετε είχαμε λάβει μια πληθώρα απαντήσεων από Υπουργεία, από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπήρξε μια γενικότερη, ευρύτερη συμφωνία ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εφιστάμενο πλαίσιο και να μην αλλάξει τίποτα. Μετά την απόφαση λοιπόν αυτή, την οποία θεωρώ σωστή απόφαση, οφείλουμε να δράσουμε εντός αυτού του πλαισίου. Ο έλεγχος καταλληλότητας λοιπόν έδειξε ότι χρειάζεται καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, έτσι ώστε να προστατεύει καλύτερα η φύση και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Το αποτέλεσμα λοιπόν του ελέγχου καταλληλότητας ήταν ότι χρειάζεται να αυξηθεί η προστασία. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε το σχέδιο δράσης, το οποίο, όπως ανέφερα στην ομιλία μου, ε, είναι ένα σχέδιο για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον και την οικονομία. Συζητήθηκε και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι και η οδηγία και το σχέδιο δράσης έχουν στόχο να βελτιώσουν την εφαρμογή και να ενισχύσουν την προστασία των ειδών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ε, παρερμηνεύονται όπως μας συμφέρει. Και από τα σχόλιά σας συμπεραίνω ότι ένα από τα αποτελέσματα των δράσεών μας ήταν να, ανακτήσει, να ανακτήσουν κάποια είδη τον πληθυσμό τους σε ορισμένες περιοχές. Όμως, οι οδηγίες αναφέρονται σε 1500 είδη. Και σίγουρα υπήρξαν κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά έχουμε και πολλά αρνητικά αποτελέσματα σε ό,τι φορά την ανάκτηση της βιοποικιλότητας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Νομίζω ότι το ζήτημα του λύκου είναι ένα θέμα που το συζητώ τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, με διάφορους, με βουλευτές, με όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς. η ανάκαμψη του πληθυσμού του λύκου έχει άμεσες επιπτώσεις με τη γεωργία. Έτσι λένε. Όμως, εγώ δεν, εμένα δεν με πανικοβάλλει αυτό. Με πανικοβάλλουν οι επιπτώσεις της ε, γεωργίας στα υπόλοιπα 1499 είδη. Γι' αυτό λοιπόν πάντα πιστεύω πως είναι χρήσιμο να συζητάμε τις λύσεις. Για τους λύκους θα αναφερθώ στη συνέχεια και για τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά να πω πρώτα ότι πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το γενικότερο ζήτημα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχει προκύψει ανάμεσα στην ε, παρουσία των ζώων σε περιοχές όπου υπάρχει εκτεταμένη γεωργία και κτηνοτροφία. Πάντα το έλεγα και θα συνεχίσω να το λέω. Νομίζω πως το, η σύγκρουση δεν είναι ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, αλλά ανάμεσα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους αγρότες, ανάμεσα στις ε, τοπικές και τις εθνικές αρχές, στα κράτη-μέλη και τις Βρυξέλλες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολύ συχνά αυτές ακριβώς οι συγκρούσεις είναι εκείνες που μπαίνουν εμπόδια στις ε, λύσεις που ψάχνουμε να βρούμε. Και κάτι άλλο. Ε, το θέμα εδώ είναι αν πρόκειται για κάτι αδύνατο ή για κάτι εφικτό. Νομίζω πως πρέπει όλα να τα εξετάζουμε στο κατάλληλο πλαίσιο, να μιλήσουμε για συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μας ε, Γίνεται λόγος για τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων ζώων σε πρόβατα. Αυτό εντάξει δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, είναι γεγονός. Όμως πρώτα οφείλετε να καταλάβετε ότι το θέμα εδώ είναι εάν η κατάσταση αυτή είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Γι' αυτό, να σας δώσω μερικά στοιχεία. Ε, τα πρόβατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 30 χρόνια μειώθηκαν από 136 εκατομμύρια σε 86 εκατομμύρια μέσα σε 30 χρόνια. Μειώθηκε ο αριθμός των προβάτων και η απώλεια ήταν της τάξης του 1,6 εκατομμυρίου προβάτων κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα πρόβατα που χάνονται από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων ζώων είναι 20.000. 20.000 από τα 86 εκατομμύρια. Μιλάμε για 0,02%. Δεν λέω ότι επειδή το ποσοστό είναι τόσο μικρό, σχεδόν αμεληταίο, δεν πρέπει να το εξετάσουμε καθόλου, αλλά να κρατήσουμε μία αναλογικότητα. Διότι το ε, υπόλοιπο από τα 1,6 εκατομμύρια πρόβατα που πεθαίνουν κάθε χρόνο ε, οφείλεται σε άλλες αιτίε, σε ασθένειες, σε, άλλου είδους απώλειες. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, ας μιλήσουμε για το λύκο και τα πρόβατα, αλλά ας ε, δούμε και πόσο διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση. Ας μην πανικοβαλόμαστε λοιπόν, να βρούμε τη λύση. Μετά, Θεωρώ πως τα κράτη-μέλη έχουν απεριόριστες ε, δυνατότητες δράσης, μπορούν να βρουν λύσεις ε, τοπικά. Προσωπικά εγώ, το επιτελείο μου, η υπηρεσία μου, όλοι οι συνεργάτες στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, επενδύσαμε πάρα πολύ χρόνο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες, με εκπροσώπους της πολιτικής έτσι ώστε να βρούμε αυτές τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις όμως είναι για τοπικά ζητήματα. Και τα προβλήματα διαφέρουν από μέρος σε μέρος. Γι' αυτό λοιπόν οι λύσεις πρέπει να είναι και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες του, της κάθε περιοχής. Δεν γίνεται από τις Βρυξέλλες να βρούμε τη μαγική λύση που θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Διότι υπάρχουν διαφορές. Μετά, Ορισμένες φορές, ορισμένα κρατημέλη υπερθεματίζουν ε, την οδηγία. Γι' αυτό λοιπόν στην ομιλία μου είπα ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν σχέδια διαχείρισης, ε, λύσεις, τα οποία θα συμμορφώνονται όχι μόνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και με την εθνική, διότι δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε για λύση Γιατί πολύ εύκολα μία λύση που θα προτείνουμε εμείς θα σκοντάψει στα εθνικά δικαστήρια. Και πολλές φορές τα δικαστήρια είναι αυτά που δίνουν δίκιο στα κράτη. Ε, σίγουρα είμαι υπέρ των λύσεων σε τοπικό επίπεδο, όμως ε, με ενοχλεί αρκετά ότι, το, το, ότι πολλές ε, περιφέρειες, πολλά κράτη προτιμούν να αποφεύγουν τις ευθύνες τους και να πετάνε τον μπαλάκι πάλι στις Βρυξέλλες. Τέλος, να πω ότι ανέφερα ήδη πως τα μέτρα διαχείρισης είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να ανακάμψουν, να ανακάμψει ο πληθυσμό ε, του λύκου. Ο πληθυσμό των ειδών. Ακριβώ διότι σε πολλές περιοχές ο πληθυσμός των λύκων βρίσκεται σε μη βιώσιμα επίπεδα ακόμα, σε ελάχιστες περιοχές ο λύκος έχει αυξηθεί σε πληθυσμό ώστε να ξεπεράσει το κατόφλι της βιωσιμότητας. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε φορά που συζητώ με κάποιον σχετικά με το θέμα αυτό, τους λέω ότι αν καταφέρετε να με πείσετε με επιστημονικά στοιχεία όχι να μου δείχνετε μια φωτογραφία από ένα πρόβατο που έχει σκοτώσει λύκο. ένα από τα 1,6 εκατομμύρια που χάνονται κάθε χρόνο. Αν καταφέρετε λοιπόν να μου αποδείξετε με στοιχεία ε, ότι γι' αυτό ευθύνατε, τότε θα σα πιστέψω. Αν ψάχνετε και ζητάτε από μένα λευκή επιταγή για να εξαφανίσουμε όλου του λύκου, δεν πρόκειται, ξεχάστε το, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εκεί όπου οι πληθυσμοί των λύκων βρίσκονται κάτω από τα ανεκτά επίπεδα, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να ανακάψει το είδος στις περιοχές εκείνες, όπου μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι λύκοι έχουν αυξηθεί πάνω από το κατόφλι αυτό τότε εντάξει ας βρούμε ένα σχέδιο διαχείρισης ε, του πληθυσμού. και ας περάσουμε από, την μία, από το ένα στάδιο στο άλλο, από το πώς να αυξήσουμε τον πληθυσμό στο πώς να τον διαχειριστούμε καλύτερα. Δεν έχει υποβληθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο μέχρι τώρα και αυτό επιβεβαιώνουν τις υποψίες μου. Είτε μιλώ με κυνηγού, είτε μιλώ με κτηνοτρόφους, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω. Τους ρωτάω κάθε φορά, με τι ιδιότητα μου μιλάτε, ως κυνηγό, ως κτηνοκτρόφος, για να σας απαντήσω καταλήλως. Πιστεύω ότι το κάθε σχέδιο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ε, κάθε περιοχής. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες έχουν χορηγηθεί εξαιρεσει και έχουμε εγκρίνει ε, σχέδια, όπως νομίζω στη Γαλλία, σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, αλλά δεν μπορούμε και πάλι να πάρουμε το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, γιατί ακόμα και μέσα στην ίδια χώρα υπάρχουν διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Διάβασα τη μελέτη που έγινε για λογαριασμό της Επιτροπής Γεωργίας σχετικά με την αύξηση του πληθυσμού ε, του λύκου και η μελέτη στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε. Σε αυτό που λέμε δηλαδή τόση ώρα. Τώρα, σχετικά με τα πουλιά. Παρότι τα μέτρα είχαν θετικές ε, επιπτώσεις, έχουμε αρνητικό ε, ισολογισμό. Το 60% των πουλιών και εξίσου μεγάλο ε, ποσοστό διατημάτων βρίσκονται σε ύφεση. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μείωσης του αριθμού και των ειδών των πουλιών, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε. Θέλουμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες αιτίες ή να τις δούμε όλες συνολικά. Η μείωση του αριθμού των ε, πουλιών και των ειδών των πουλιών οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Και ακριβώς επειδή το πρόβλημα προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, τότε μπορούμε, επειδή είμαστε άνθρωποι, να το λύσουμε. Ε, ξεκινώντας από τις ε, γεωργικές πρακτικές, είχαμε τις ε, σχετικές εκθέσεις για την κατάσταση της ε, φύσης, της γης, είχαμε την ενδιάμεση αξιολόγηση τη στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα. Όλα αυτά Όλες αυτές οι μελέτες μας έδειχναν ότι τα αίτια είναι τα ίδια και αυτό που δεν αναφέρεται λοιπόν εδώ, αυτό που δεν συζητάμε είναι τις συνέπειες της γεωργίας. Υπάρχουν, υπάρχει καλή, υπάρχουν καλές γεωργικές πρακτικές και κακές γεωργικές πρακτικές και πρέπει, θεωρώ, ε, η λύση να είναι απλή. Να στηρίζουμε τις ε, καλές πρακτικές και να ε, σταματήσουν οι κακές γεωργικές πρακτικές. Μιλάω για τα ζυζανιοκτώνα, για τα φυτοφάρμακα, η βιοπικιλότητα. Επίσης, να σας πω ότι δεν αφορά μόνο την ξηρά αλλά και τη θάλασσα. Υπάρχει στρατηγική για τα πλαστικά στις θάλασσες. Τα πλαστικά είναι η μεγαλύτερη πληγή των ωκεανών. Όμως, σε σχέση με το πρόβλημα για τις θρεπτικές ουσίες, ε, τα πλαστικά δεν είναι τίποτα. Η έλλειψη θρεπτικών συστατικών προκαλεί άπειρες φορές περισσότερη βλάβη στους ωκεανούς από τα πλαστικά. Και ο τρόπος που χειριζόμαστε το θέμα με τα πλαστικά θα καθορίσει, λέτε, το μέλλον των ωκεανών. Διαφωνώ, διότι ξεχνάμε και άλλα, τα άλλα προβλήματα, τις αλλαγές των, ε, ε, στα οικοσυστήματα, την επιδείνωση των οικοσυστημάτων, την αποψήλωση των δασών. Σίγουρα το κυνήγι επίσης ευθύνεται εν μέρη για την επιδείνωση της κατάστασης. Το κυνήγι όμως μπορεί να γίνει με τρόπο βιώσιμο. Επίσης, η μείωση των ειδών και του αριθμού των πτηνών είναι επίσης κάτι ανησυχητικό. Γίνεται λόγος για τα μεταναστευτικά πτηνά, όμως πρέπει να συζητήσουμε για όλα, διότι μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ε, πτηνών, όχι μόνο τα μεταναστευτικά. Επίσης, είπαμε ότι έχουμε συμφωνήσει πως η οδηγία για τα πουλιά είναι κατάλληλη, εξακολουθεί να είναι κατάλληλη. Όμως, είναι κατάλληλη μόνο εφόσον εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει νόημα να θεωρούμε μια οδηγία κατάλληλη την οποία δεν εφαρμόζουμε. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλουμε μια γενικότερη προσέγγιση διότι διαφορετικά, αν λειτουργούμε επιλεκτικά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη βιοπικιλότητα, τη απώλεια βιοπικιλότητας, τα πτηνά, θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους. Και αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πτηνά και από την ανθρώπινη δραστηριότητα, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι πολιτικές μας ε, δρουν προς όφελος της φύσης και όχι εναντίον της. Γι' αυτό ο συνάδελφός μου, ο Φιλ Χόγκαν και εγώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Έχουμε μια ευκαιρία μέσω της ε, οδηγίας αυτής, γι' αυτό λοιπόν και θέλω να είμαι σίγουρος ότι ε, στην κοινή γεωργική πολιτική θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα αποδώσουν καρπούς. Τώρα, συγκεκριμένα για τη Μάλτα. Πρόκειται για κάτι το οποίο υπερβάλλεται κατά τη γνώμη μου. Να μιλήσω για τις παραβάσεις στη Μάλτα. Είχε για κάποιες παγίδες σπίνων και θα μπορούσαμε να έχουμε σταματήσει αυτή τη διαδικασία διότι η Μάλτα απέσυρε την ε, παρέκκληση αυτή τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε κλείσει το θέμα, απλά για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξανανοίξει αυτή η πρακτική την επόμενη σεζόν όσον αφορά τα ορτίκια και τις 18 στη Μάλτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβήτησε την παρέκκληση αυτή Πήγαμε στο δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της Μάλτας όσον αφορά τις 18 και τα ορτίκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο λοιπόν. Αυτό που κάναμε όμως, διότι υπήρχε μια προϋπόθεση στην απόφαση αυτή, η παρέκκληση να σταματήσει μόλις ε, αλλάξει το καθεστώς των πτηνών. Μόλις ε, θεωρήθηκε ευάλωτος ο πληθυσμός σε 18 ώρες, ε, ξεκίνησαν μέτρα. Η Μάλτα ξεκίνησε μορατόριουμ το 2016 για το κυνηγητή ώρας. Και για να σας καθησυχάσω όλους, για μένα υπήρχε το θέμα της δεκαυτούρας στη Μάλτα που ανέρχεται σε περίπου 2.000 άτομα και την Ισπανία και το υπόλοιπο της Ευρώπης 2,4 εκατομμύρια. Και εγώ είπα, εγώ θέλω να σταματήσω το κυνήγι την άνοιξη στη Μάλτα και το κυνήγι το φθινόπωρο σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχει νόημα να σκοτώνουμε προστατευόμενο είδες, είτε αυτό γίνεται στην Ισπανία είτε γίνεται στο Βορρά. Η Μάλτα εφήρμοσε μορατόριουμ και αν ε, μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη εφαρμοζόταν σχέδιο για την 18 τότε εντάξει, αλλά δυστυχώς ε, τα κράτη-μέλη δεν το δέχτηκαν αυτό. Ναι, σωστά σταματήσαμε τη Μάλτα, αλλά σώσαμε τη 18 Τη στιγμή που θα θανατώνονται 2,4 εκατομμύρια στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Γι' αυτό πάντα λέω, ας κοιτάξουμε την ευρύτερη εικόνα. Διότι θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η κυρία Σράια Πύρικ. Όσον αφορά τους κορμοράνους ε, και τα δύο είδη χήνας που αναφέρατε, για τα οποία έχουν ζητήσει παρεκκλήσει τα περισσότερα κράτη-μέλη, και τα τρία αυτά πτηνά βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη και μάλιστα ανάλογα από το αν μετρήσουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα. Όλα εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα τροφής. Όσον αφορά τους κορμοράνους, μπορώ να σας πω ότι το Βέλγιο, η Ιδανία, η Εστονία, η Φιλανδία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Λιθουανία, οι κάτω χώρες, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν παρεκκλήσεις. Το να έχουμε λοιπόν πάντα παρεκκλήσεις ε, δεν έχει νόημα. Αν οι παρεκκλήσεις ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες και με την εθνική νομοθεσία, τότε εάν δεν αποτελούν απλά δικαιολογία για να σκοτώνουμε τα ζώα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμόζονται οι παρεκκλήσεις. Η κυρία Μελιόρ δύο πράγματα ρώτησε. Πρώτον, όσον αφορά τα δεδομένα, την επιβολή δεδομένων για το λύκο. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν μία προθεσμία από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα, αξιολογούνται από την EAA και από τη δική μας Γενική Διεύθυνση. Όσον αφορά τις άλλες ερωτήσεις. Νομίζω ότι σε αυτές θα πρέπει να απαντήσει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι μέχρι να δημοσιευτεί η αξιολόγηση, νομίζω θα υπάρχει άλλος επίτροπος. Όσον αφορά το ποια θα είναι η θέση των Ελβετών ε, στην επόμενη σύμβαση της Βέρνης, μπορώ να σας πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση για την σύμβαση της Βέρνης, η Ελβετία είπε ότι θέλει να επανέλθει στις προτινόμενες τροπολογίες για τον Λύκο σε μεταγενέστερη συνεδρίαση που θα έχουν εξεταστεί τα συμπεράσματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η θέση της Ελβετίας. Η κυρία Γκροστέτ ανέφερε τη Γαλλία και τα προβλήματα με το Λύκο. Συμφωνώ απολύτω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά προτείνουμε λύσεις. Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να τις εφαρμόσουν. Δεν θα πρέπει να μας ε, θεωρήσετε υπεύθυνους για τη μη εφαρμογή αυτών των λύσεων. Μπορεί να πω κάτι με το οποίο διαφωνείτε. Εγώ θα το πω όμως. Πολιτικός είμαι όπως και εσείς. 38 χρόνια ήμουνα στο κοινοβούλιο. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι η ψήφοι. Εάν οι υπουργοί, οι πολιτικοί, τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι πρέπει να λάβουν απόφαση που μπορεί να είναι δημοφιλής στους μεν, όχι όμως στους δε, μπορεί να κερδίσουμε ψήφους από εδώ, να χάσουμε από εκεί όμως, τότε υπάρχει μόνο μία λύση, να κατηγορεί κανείς τις Βρυξέλλες. Αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Και το επαναλαμβάνω εδώ, διότι το έχω πει σε όλους όσοι λένε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά. Τα αντιμετωπίζουμε και με το παραπάνω. Ε, νομίζω ότι ο κύριος ε, τώρα έχει να, πρέπει να φύγει, αλλά συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει. πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της αστικοποίησης. Γνωρίζουμε ότι κάποια χρονική στιγμή οι λύκοι δεν πλησίαζαν όταν άκουγαν θόρυβο, όταν έβλεπαν φως. Τώρα νομίζω ότι εξοικειώνονται σιγά σιγά. Πρέπει να βρούμε λοιπόν σχετικές λύσεις. Όπως είπα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία συζήτησα το θέμα, το θέμα του λύκου. Είναι τελείως διαφορετικό το πρόβλημα της Σουηδίας όμως. Εκεί δεν έχει μόνο να κάνει με τους αριθμούς, έχει να κάνει με τις γενετικές ασθένειες που έχουν αναπτύξει οι λύκοι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν λοιπόν μόνο τα νούμερα. Μας ενδιαφέρει και το αν συνδέονται με άλλα προβλήματα οι λύκοι, όπως είναι κάποιες ασθένειες. Κύριε Χόισλινγκ, ναι, μιλάμε για την απώλεια βιοπικιλότητας. Είναι ατυχές το ότι δεν είναι θέμα απώλειας ε, τη μια χρονιά σε σχέση με την προηγούμενη, είναι μια γενική τάση. Ναι, είναι επίγον το θέμα. Δύο προβλήματα έχουμε αυτά που βλέπω γύρω μας. Πρώτον, απώλεια της βιοπικιλότητας. Συμβαίνει και αποτελεί πρόβλημα. Για μένα όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι γίνεται με τέτοια ραγδαία ταχύτητα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο επίγον είναι το θέμα αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα όταν μιλάμε για τη βιοπικιλότητα. Πάντα Δίνω το ίδιο παράδειγμα ε, σχετικά με την ε, κοραλιογενή ατόλη ε, στην Αυστραλία, το Great Barrier Reef. Πριν κάποια χρόνια τέθηκε το ερώτημα αν θα μπορέσει να αντέξει στην αλλαγή του κλίματος. Πέντε χρόνια μετά κάποιος επιστήμονας προσπάθησε να απαντήσει και κατέληξε σε αρνητική απάντηση. Δεν θα μπορέσει να αντέξει τα αποτελέσματα της ε, αλλαγής του κλίματος ε, και τα αποτελέσματα θα τα δούμε το 2050. Πέρσι όμως το μισό αυτής της ατόλης είχε ε, πεθάνει. 20 χρόνια πριν από την ημερομηνία που μας έδωσαν οι επιστήμονες. Δεν είναι λοιπόν μόνο το τι συμβαίνει, είναι και το ότι όλα αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι επιστήμονες. Και παρόλα αυτά πάντα συζητάμε το θέμα, μιλάμε για τα επιμέρους μέτρα που θέλουμε να λάβουμε, μιλάμε για τις μικρές αιτίες, διότι δεν έχουμε το θάρρος να αντισταθούμε στα μεγάλα λόμπι και να πούμε να, ορίστε, αυτά προκαλείται. Έτσι συμβάλλεται στην ε, απώλεια της, της ε, βιοπικιλότητας. Ε, και όχι μόνο δημιουργείτε προβλήματα, αλλά σας επιχορηγούμε κιόλα. δίνω το 1 τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μολύνουμε το περιβάλλον και, και μετά πληρώνουμε άλλα τόσα για να, για να διορθώσουμε την κατάσταση. με την κοινή γεωργική πολιτική θέλουμε να βεβαιωθούμε όλοι οι πόροι να δίδονται για να προστατεύσουμε τη φύση και όχι το ανάποδο. Μπορεί να μην γίνομαι πολύ δημοφιλής όταν τα λέω αυτά, αλλά νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα λέω. Η κυρία Εύη. Δεν ξέρω που κάθεται. Είπατε ότι οι παρεκκλήσεις δεν εφαρμόζονται σωστά. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος παρακολουθεί από κοντά όλα τα μέτρα. Δεν ε, θέλω να περηφανευτώ για τη στατιστική μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό ε, διαδικασιών επί που συνδέονται με την φύση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς ε, να κατηγορήσει την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και ότι δεν παρακολουθεί την κατάσταση. Η δημόσια ασφάλεια είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε, συμφωνώ. Κύριε Ντόρφμαν. Ναι, Πράγματι έχετε δίκιο για την Κροατία, γι' αυτό ανέφερα ότι συνεχώς ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές, συνεχώς ανταλλάσσουμε λύσεις και κάτι που κάναμε και το οποίο δεν διαχειρίστηκε μόνο, αλλά πλήρωσε και όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν η δημιουργία της μεγάλης πλατφόρμας σαρκοβόρων. Όχι μόνο δημιουργήσαμε την πλατφόρμα, δημιουργήσαμε και μια σειρά άλλων πλατφορμών σε διάφορα κράτη-μέλη και σε διάφορες περιφέρειες. Νομίζω ότι έτσι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητάμε, να έχουμε ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερομένους. Και δεν καταλαβαίνω. Τα κάνουμε όλα αυτά για να στηρίξουμε τη γεωργία και από αυτές τις πλατφόρμες σαρκοβόρων υπάρχουν ε, εκπρόσωποι των γεωργών που δεν θέλουν να συμμετέχουν. Πώς να το εξηγήσω εγώ αυτό στους άλλους ενδιαφερομένους. Οι εκπρόσωποι των γεωργών λένε ότι α, δεν μας ενδιαφέρει η συμμετοχή σε αυτές τις πλατφόρμες. Επαναλαμβάνω, λυπάμαι πολύ που τα λέω όλα αυτά. Ξέρω ότι είσαστε πολύ ειλικρινείς όπως ε, και εγώ, αλλά κάποια από αυτά τα πράγματα δεν βγάζουν νόημα κατά τη γνώμη μου. Ο κ. Σπρέναν ανέφερε ότι μπορεί να χρειαστεί να κοιτάξουμε την έρευνα και τα ωφέλη από αυτήν. Ναι, πράγματι, η λύκη είναι τμήμα του οικοσυστήματος και επιφέρουν ωφέλη στο οικοσύστημα. Θεωρούμε τα μεγάλα σαρκοβόρα ζώα μόνο κάτι αρνητικό, αλλά συμβάλλουν σημαντικά στα οικοσυστήματα. Εάν υπάρχουν έρευνες που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τα ωφέλη των λύκων και των άλλων μεγάλων σαρκοβόρων, νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε διάφορες ερωτήσεις. Okay, thank you very much. Uh, λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Επίτροπο. Είχαμε πολλές ερωτήσεις. Ε. Είχαμε βέβαια προγραμματίσει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε που καθίσατε μαζί μας περισσότερο χρόνο από όσο είχατε αρχικά προγραμματίσει και θα παρακολουθήσουμε μαζί σας ε, την κατάσταση αυτή και την εξέλιξή της στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Chair, can I make a point of order, please? Ένα διαδικαστικό, Πρόεδρε, αφού φύγει ο Επίτροπος, αν θέλετε. Point of order. Which... On this? No. A point of... Yes, uh, please. Κύριε Γκερμπράντι. Ναι, Πρόεδρε, ε, πιστεύω ότι η κατανομή του χρόνου ομιλίας δεν ήταν δίκαια. Δώσατε το λόγο στους S&D και στους ELK με τέσσερις ομιλητές, πέραν των οποίων Τρει ομιλητέ ζήτησαν το λόγο. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι θα έχουμε μόνο ένα γύρο, έτσι όπως τον κατανείματε. Ήθελα να το πω αυτό, δεν θα αλλάξει τίποτα βέβαια, αλλά πιστεύω πραγματικά και θέλω να καταγραφεί δεν ήταν δίκαιο. Ε, ο κατάλογος των ομιλητών έπρεπε να έχει γίνει γνωστός από τους ε, συντονιστές. Είχατε έναν ομιλητή ζητήσει. Εγώ συνήθως ε, δίνω τον λόγο στους ομιλητές που ζήτησαν. Σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη περίπτωση ότι δεν είχαμε χρόνο, λέει η Πρόεδρος. Θα πάμε τώρα στο, στα πορίσματα του ICIJ, των ε, του διεθνούς αυτού, της διεθνούς ομάδος ε, δημοσιογράφων σχετικά με τους φακέλους για τα εμφυτεύματα λοιπόν. Ε, θέμα για το οποίο έχουμε εκπροσώπους του ICIJ των δημοσιογράφων δηλαδή έρευνας, τον κύριο Σάιμον Μπάουερς που είναι Ευρωπαίος συντονιστής. Έχουμε τον CEO της Metac Ευρώπη και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Growth, κύριο Πέλτομάκη. η έκδοση ελωτοματικών ή ψευδός, εμπασχελτώσει πλαστών εμφυτευμάτων έχει βρει το δρόμο της προς τον τύπο σε διάφορες χώρες. Ο τομέας έχει μια πολύ υψηλή αξία και έχει παρακολουθηθεί επί χρόνια σχετικά με τα συστήματα που πρέπει να διέπουν τη ρύθμισή του την ομοθετική και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ως επικεφαλής επιτροπή, ως αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα και πολύ με μεγάλη ικανοποίηση σημειώνω ότι έχουμε αυτήν την ε, ανταλλαγή σήμερα και καθότι έχουμε ήδη αργήσει δεν θα μακρηγορήσω άλλο και θα καλέσω καταρχάς ε, τον κύριο Bowers να λάβει το λόγο για 10 λεπτά το πολύ αν θέλετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που καλέσατε το ICIJ να μιλήσει στην Επιτροπή σας. Η φάκελη των εμφυτευμάτων ήταν ένα έργο το οποίο συντονίσαμε ως ICIJ που είναι μια σύμπραξη ενώσεων δημοσιογράφων παγκόσμιας εμβέλειας στην Ευρώπη αφορά περί τους 100 δημοσιογράφους σε 30 διαφορετικά μέσα 16 διαφορετικών χωρών. Θα βάλω στην ε, οθόνη κάποια από τα μέσα που συνεργάζονται. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν ως ομάδα και συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να εξιστορήσουμε θέματα τα οποία δεν μπορούμε από μόνοι μας ή σε μια σκοπιά μιας και μόνο χώρας. Μια Ολλανδή δημοσιογράφος το 2014 αγόρασε μια τσάντα μανταρινιών και τα μοίρασε ως εμφυτεύματα για γυναίκες για, για την θεραπεία της ακράτειας. Επί του επεισοδίου αυτού οικοδομήθηκε ένας φάκελος τεχνικός, ο οποίος διαβιβάστηκε σε διάφορους αρμόδιους οργανισμούς ε, πιστοποίησης. Κανείς από τους οποίους δεν εσημείωσε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όλοι προσυπέγραψαν τον τεχνικό φάκελο, τον τεχνικό εντό εισαγωγικών. Ε, η δημοσιογράφος δεν σταμάτησε αυτή, θεώρησε ότι το πρόβλημα ήταν ευρύτερο, πιο σημαντικό και ήρθε στην, στο ICIJ, εμείς αναπτύξαμε ένα δίκτυο συνεργασίας και αναδείξαμε το θέμα. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω επίσης ε, τρεις ασθενείς και ίσως με την ευκαιρία να δείξουμε κάποια από τα θέματα που έχουμε καλύψει. Είναι αδύνατο να καλύψουμε όλα τα ευρήματα. Η πρώτη ασθενής είναι πάνω αριστερά. Είναι η Maureen Μακλίβ από το Λονδίνο και αυτή είναι η δική της ιστορία. είναι πρώτη από δύο διαφάνειες, με πριν και μετά αν θέλετε. Ξεκινάει πολύ αισιόδοξα η προσωπική της ιστορία. Είναι η πρώτη ασθενής που λαμβάνει έναν ε, βηματοδότη ο οποίος δεν είχε καλώδια που ε, τον συνέδε με την καρδιά. Αυτός ήταν χωρίς καλώδια και συνδεόταν απευθεία επειδή ήταν πάρα πολύ μικρός, και συνδεόταν απευθεία στην καρδιά, καθότι τα καλώδια πολύ συχνά ήταν συνδεδεμένα με περιπλοκές τη υγεία. Ε, αρχικά η κυρία αυτή έλεγε ότι αισθάνεται σαν καινούριο άνθρωπος, χωρίς ακροδέκτες λοιπόν, Ο Dan Στάρξ, ο οποίος υπήρξε ο, ε, ο υπεύθυνος της επιχείρησης που ε, παρήγαγε το NanoSteam, αυτό το συγκεκριμένο βηματοδότη, είχε ε, εμφανιστεί στη τηλεόραση για να παρουσιάσει τα επιτεύγματα αυτού του νέου τεχνάσματος και έλεγε είμαστε οι πρώτοι που το πετυχαίνουμε, πρόκειται για μια, ένα τεράστιο βήμα, μια τεράστια πρόοδο και είμαστε ηγέτες πλέον του πεδίου κτλ. Αυτή τώρα είναι, που θα δείτε είναι η επόμενη διαφάνεια, όπου έχει αλλάξει η εικόνα μετά από λίγα χρόνια, με μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Ο κύριος Στάρξ είχε πει στην τηλεόραση ότι ο βηματοδότης Μωρίν θα κρατούσε για 19 χρόνια, κράτησε 3 η μπαταρία του οποίου ε, πολύ γρήγορα έπαψε να λειτουργεί και σε άλλους ασθενείς, πολλοί άριθμους άλλους ασθενείς. που χρειάστηκε να τους αλλάξουν την μπαταρία και ήταν μια απλή αλλαγή σε αρκετέ περιπτώσει, αλλά όχι στην περίπτωση της Μωρήν που χρειάστηκε να χειρουργηθεί και πάλι. Χρειάστηκε λοιπόν να υποστεί νέα εγχειρητική διαδικασία που δεν περίμενε ποτέ, ώστε να τις ε, τοποθετηθεί, να, σε, να τις εμφυτευτεί παραδοσιακός βηματοδότης. Ε, δήλωσε λοιπόν ότι αισθάνθηκε ότι τη μεταχειρίστηκαν σαν σκουπίδι. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το έλεγε αυτό. Αν ήσασταν εσείς στη θέση της, θα ήταν λογικό να ρωτήσετε τι δοκιμές έκανε η NanoSteam. Τι δοκιμές έκαναν για το προϊόν αυτό. Η απάντηση είναι 33 δοκιμές ανθρώπινες και 30 επί προβάτων. Μετά από αυτόν ακριβώς τον αριθμό δοκιμών πιστοποιήθηκε ως ε, επαρκές για τη δημόσια υγεία. Το νάνο είναι ένα από πάρα πολλά προϊόντα. Οι ιατροτεχνικές συσκευέ οι οποίες διέρχονται πολύ ελλειπών δοκιμών και τεστ Και αυτό οφείλεται στην ελλειπή και εξαιρετικά ελαφρά νομοθεσία. Και ε, κυρίως έλλειψη κυρώσεων σχετικά με ε, ε, βλάβες που μπορούν να έχουν οι ασθενείς. Άλλη μια περίπτωση είναι η Ζακλίν Ρούς, η οποία αποφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε εμφύτευμα μαστού, έχει υποφέρει από ε, χρόνια αλγία, ε, έχει υποβληθεί σε μια σειρά από εγχειρήσει. Ε, της είπαν ότι αυτό είχε σχέση με την ψυχική της υγεία. Αυτή τους είχε προτείνει ότι μήπως όλα αυτά σχετίζονταν με τα εμφυτεύματα σιλικόνης που είχε στον μαστό. Της είπαν ότι έλεγε ανοησίες έως ότου επέμεινε να ελέγξουν τον ιστό μετά από κάποια εγχείρηση και βρήκαν ότι πραγματικά είχε επίπεδα σιλικόνης που δεν έπρεπε να βρίσκονται στον οργανισμό. Τα εμφανιτέματα μαστού είναι μαζί μας από δεκαετία του 60. Δεν είναι κάποιο καινούριο προϊόν όμως των nanosteam. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε επικαιροποιημένες ενδείξεις σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι γυναίκες που προχωρούν σε τέτοιου είδους εγχειρήσεις, επεμβάσεις. Αυτό είχε τεθεί πριν από δεκαετίες σε κάθε πιθανό ευρωπαϊκό θεσμό από σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Ο τελευταίος ασθενής στον οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ανώνυμος, δεν έχουμε όνομα, είναι πολύ πρόσφατη περίπτωση του Ιανουαρίου όπου η Medtronic ανακάλεσε άνω των 150.000 βηματοδότες και εδώ έχουμε μία ανώνυμη αναφορά ενός ασθενούς από το Ipswich στην Αγγλία που είπε στην τοπική του εφημερίδα και μετά από επιστολή του γιατρού του ότι κάποια πράγματα που έλεγαν στην επιστολή με ανησύχησαν Ιδιαίτερα όταν είπαν ότι κανείς ακόμα δεν έχει πεθάνει. Μου φάνηκε περίεργο να λένε κάτι τέτοιο. Εξεπλάγιν, λέει ο ανώνυμος ασθενής. Και ανησύχησα. Και η συγκρατημένη γλώσσα που χρησιμοποιεί εκεί αντιλαμβάνεται κανείς πώς θα πρέπει να αισθάνεται κανείς όταν έχει διαβάσει ένα τέτοιο νέο. Η Μετρόνικ στην ανακοίνωση προς τους γιατρούς έλεγε ότι είχε τέσσερις περιπτώσεις, τέσσερα κρούσματα διακοπής της όθησης ε, λόγω λάθους ηλεκτρικού κυκλώματος μέσα στον βηματοδότη. Αλλά η πραγματική ερώτηση είναι πόσες περιπτώσεις έχει η Μετρόνικ, πώς μπορεί να ξέρει ότι υπάρχουν μόνο τέσσερις Δηλαδή αν έχει εντοπίσει ανεφοβολία τέσσερι, τέσσερις, πόσα ερωτηματικά γύρονται για πόσους άλλους βηματοδότε που είναι εμφυτευμένοι σε ασθενείς. Και ήθελα να προσπαθήσετε να φανταστείτε ότι είστε αυτός ο άνθρωπος που έχει λάβει την επιστολή σχετικά με την ανάκληση αυτού του βηματοδότη. Τι θέλετε να μάθετε. Ακούτε στη φωνή του την τραγική ερώτηση μήπως υπάρχει περίπτωση να πεθανώ. Και η επιστολή δεν φαίνεται να τον καθιστά σαφές. Η επιστολή λέει δεν πέθανε κανείς ακόμα. Αν ήσασταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα είχε ε, κατηγοριοποιηθεί ως ανάκληση κατηγορίας 1, λόγω σοβαρότητα της ανησυχίας δηλαδή συμπεριλαμβανομένης απειλής θανάτου στην Ευρώπη, τι άλλο θέλετε να ξέρετε. Τι δοκιμές ασφαλείας έχουν γίνει επί των βηματοδοτών αυτών. Πόσες ενδείξεις είχαμε ότι μπορεί και κάτι να πάει στραβά με το προϊόν αυτό, με την συσκευή αυτή. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει τουλάχιστον μια διαφάνεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καμία. Στις Ηνωμένε Πολιτείε μπορεί να διαβάσει κανείς την έκθεση της FDA για σχετικές ε, αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό στην Ευρώπη μηδέν. Και αν θέλει κανείς να βρει πόσες δοκιμές, λαμβάνει απάντηση ότι που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική και καθόλου δεν επιβεβαιώνει κανέναν. Μάλιστα η τελευταία πλήρης ε, έκθεση που έχουμε σχετικά με τη συσκευή αυτή είναι του 1999. Η ημερομηνία από την οποία έγιναν άνω των 500 τροποποιήσεις στα σχετικά προϊόντα. Επομένω, οι Ευρωπαίοι πολίτε αφήνονται στο απόλυτο σκοτάδι ω προ την ενημέρωση αυτή που θα έπρεπε να έχουν. Τώρα κοιτώντας την επόμενη διαφάνεια. Η διαφάνεια υποτίθεται ότι είναι στην καρδιά της ε, νέας νομοθεσίας για τις ιατροτεχνικές συσκευέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δική μας μελέτη ότι δεν έχουμε την νέα νομοθεσία ακόμα, αλλά πού βρισκόμαστε. Στα γραφήματα αριστερά έχουμε τις, τα αυξανόμενα κρούσματα συσκευών με τις οποίες έχει υπάρξει πρόβλημα σε διάφορες χώρες. Σε συγκρίσιμες χώρες. Η τάση είναι παντού ίδια. Αύξηση των επεισοδίων. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να μάθουμε είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο κανονισμό για τις ε, ιατροτεχνικές συσκευέ σε επίπεδο διαφάνειας. Και παρότι δεν έχει πει η Κομισιόν τίποτα επίσημα, μαθαίνουμε από την Κομισιόν ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να δημοσιοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τους ασθενείς και για τους γιατρούς με τους οποίους μιλάμε. Και η Κομισιόν μας, λένε, μας λέει ότι δεν θέλει να δημοσιοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των προκλινικών τεστ για αντίστοιχα δηλαδή φαρμακοτεχνικά προϊόντα. μια στάση η οποία δεν καλύπτει τον, τους επαγγελματίες του κλάδου. Επομένως, αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που μπορεί να μην αρέσει ως προς τη διαφάνεια, λέει ο μιλητής. Και η Κομισιόν μας λέει ότι με όλες αυτές τις εκθέσεις θα μπορούσε να ανησυχήσει το κοινό. Η διαφάνεια θα μπορούσε να ανησυχήσει το κοινό. Διακόπτει η πρόοδος η πρόεδρος, με συγχωρείτε, και λέει πρέπει να επιταχύνεται στον ομιλητή. Ο ομιλητής λέει μάλιστα πρόεδρε, θα επιταχύνω. Ότι ο κλάδος λοιπόν θα ήταν ακόμη πιο διστακτικός να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες εφόσον υπάρξει διαφάνεια. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν μια σοκαριστική απάντηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επόμενη διαφάνεια δίνει στοιχεία που δεν θα πάω σε λεπτομέρειε, αλλά είναι κάποιε από τι απαντήσει θα τις μεριαστώ μαζί σας αργότερα. Οι γιατροί οι επαγγελματίες ε, είναι εξοργισμένοι, απαιτούν διαφάνεια. Ε, κανένας ανεξάρτητος γιατρός δεν βρίσκεται που να μην είναι υπέρ της διαφάνειας θέματα αυτά. Ήθελα απλώς λοιπόν να κλείσω λέγοντας τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Έχουμε την ομοθεσία εκεί που βρίσκεται για τις φαρμακοτεχνικές συσκευέ Κάποια κράτη-μέλη ήδη αισθάνονται ότι πρέπει να αναλάβουν πρόσθετες διατάξεις με υποχρεωτικά μητρώα εμφυτευμάτων και σχετικών συσκευών. Αυτό το χαιρετίζει η επαγγελματική κοινότητα των ιατρών, αλλά οπωσδήποτε αυτό αποκλίνει, είναι αποσπασμένο από, την, από τον βασικό άξονα της νομοθετικής προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, όλοι οι επαγγελματίε με τους οποίους εμεί μιλήσαμε και είμαι βέβαιος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι λομπίστε, θα το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Όλοι μιλούν, όλοι κάνουν πεάνε υπέρ της διαφάνειας. Να λοιπόν, μια καλή ευκαιρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να μιλάει απλώς να υμνεί τη διαφάνεια, να την υπηρετεί με πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Περνασκόνη από την Τα Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε σήμερα να συμμετάσχω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να πω καταρχά ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι βασική σημασία, κρίσιμη σημασία τόσο για εμά όσο για όλου πιστεύω ως ε, βιομηχανία έχουμε ευθύνη για την υγεία των ασθενών. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, κρατάμε τις δεσμεύσεις μας για την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και που βελτιώνουν την ε, ποιότητα ζωής των ασθενών. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές, ε, του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νοσοκομεία, τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Τηρούμε λοιπόν τις ε, νομικές μας υποχρεώσεις και προσπαθούμε να παρέχουμε τις ε, καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς. Η προσοχή που δίνουμε στην ε, τεχνολογία της ιατρικής είναι πάρα πολύ σημαντική για να ταπεξέλθουμε στις ανάγκες των ασθενών. Είτε πρόκειται για εξοπλισμό, είτε για υψηλά εξειδικευμένα προϊόντα. κατά πάσα πιθανότητα όλοι γνωρίζουμε κάποιον που χρησιμοποιεί ένα, ηλεκτρο... ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Γι' αυτό η έρευνα που έγινε από το ICIG άλλαξε τα δεδομένα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι πλέον προηγμένης τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που μέχρι τώρα δεν είχαμε φανταστεί πριν από, ε, πριν από 10 χρόνια, πριν από μία γενιά ήταν αδιανόητο να χρησιμοποιήσουμε ε, την τεχνολογία στην ιατρική με τέτοιο τρόπο. Βελτιώνεται καθημερινά και συνεχόμενα η τεχνολογία στον χώρο της ιατρικής. Τόσο οι ιατροί όσο και οι ασθενείς απαιτούν διαφάνεια και ε, αυξημένη λογοδοσία σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά πληροφορίες που εμείς χρησιμοποιούμε ως, ε, και παρέχουμε ως βιομηχανία στους, ε, στο κοινό και στους δημοσιογράφους, ε, ελπίζουμε να τους βοηθήσει να κάνουν το έργο τους. Ελπίζουμε να υπάρξει βαθύτερη κατανόηση σχετικά με το τι συμβαίνει και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Κάποιες από τις ερωτήσεις ε, των δημοσιογράφων είναι εγκυρότατες, όμως ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι απαντήσεις που ε, παρέχει η βιομηχανία ή οι αρμόδιες αρχές ήταν ορισμένες φορές αρκετά περίπλοκες. Και παρότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία, νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ε, το κύριο μέλημά μα είναι η ασφάλεια των ασθενών. Τώρα θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η βιομηχανία πάντα στήριζε την ανάγκη ε, μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου. Ο κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ε, ρισικά διαφορετικό σε σχέση με ε, παλαιότερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, πρέπει να συμμορφωθούμε με ε, διαφάνεια ανεξάρτητα από τις ε, μεγάλες προσπάθειες ε, που θα χρειαστεί να καταβάλουμε για να το πράξουμε αυτό. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρία Πρόεδρε του, της Επιτροπής, θέλουμε διαφάνεια. Κάθε 20 δευτερόλεπτα εμφυτεύεται ένας βηματοδότης, ο οποίος σώζει ζωές. Κάθε χρόνο γίνονται εκατομμύρια χειρουργία τα οποία επιτρέπουν στους ασθενείς να ζήσουν ε, με αξιοπρέπεια και αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχει κίνδυνος πολλές φορές κάτι να μην πάει καλά για διάφορους λόγους. Οποιοδήποτε περιστατικό που αφορά ιατροτεχνολογικό προϊόν μας αφορά και μας ανησυχεί ε, έντονα. Παίρνουμε το θέμα στα σοβαρά και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα που έφερε στο φως το ICIJ και είμαστε πεπισμένοι ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ευρώπη θα δώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα του ICIJ. Ο νέος κανονισμός λοιπόν αλλάζει και βελτιώνει πολλές ε, πτυχές ε, της ασφάλειας των προϊόντων αυτών και η ρυθμιστική διαδικασία θα ε, απολαμβάνει πλέον ψηλότερες ασφάλεια και υψηλότερων προτύπων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σύμφωνα με τον κανονισμό θα ενισχυθεί η έγκριση ε, της αγοράς. Ο κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα επίσης ε, μεγαλώνει το πεδίο εφαρμογής. Αυξάνονται οι απαιτήσει για ε, κλινικές δοκιμές, για αποδεικτικά στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια ενός προϊόντος. Χρησιμοποιείται και η αρχή της ισοδυναμίας, ε, όμως ενισχύονται οι απαιτήσει για τους κοινοποιημένου ε, οργανισμούς. Πρέπει να είναι εγκεκριμένοι και να υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών. Επίσης, τα νέα προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορίες με επιπρόσθετους ελέγχους ή καινοτόμα προϊόντα θα πρέπει πλέον να περνούν ακόμα πιο αυστηρές διαδικασίες έγκρισης. Επίσης, η ελεγχη σε τακτά διαστήματα, τόσο στις αποθήκες όσο και στην αγορά, θα ε, αυξηθούν. Από τη στιγμή που εγκρίνεται ένα προϊόν, ο κατασκευαστής θα έχει τη συνεχόμενη υποχρέωση να συλλέγει ε, κλινικά επιστημονικά στοιχεία για την ασφάλεια των προϊόντων. Κάθε τρία με πέντε χρόνια οι κατασκευαστές θα πρέπει να ζητούν πιστοποίηση των προϊόντων τους παρέχοντας νέα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις τους. Ακριβώς όπως στην ε, φαρμακοβιομηχανία. Επίσης, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα μπορούν να ε, εντοπιστούν ως προς την προέλευσή τους. Η δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων επίσης εγγυάται περισσότερη ασφάλεια. Έτσι θα παρέχονται ακόμα περισσότερες πληροφορίες ε, στο κοινό, το οποίο θα έχει πρόσβαση σε ε, ετησίως επικαιροποιημένα στοιχεία. Επίσης, ε, φυσικά και θα γίνεται σεβαστός ο κανονισμός ε, για τα προσωπικά δεδομένα. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσουμε μία σφαιρική κατανόηση σχετικά με την ασφάλεια των υδροτεχνολογικών ε, προϊόντων. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν προκλήσεις ως προς την εφαρμογή του κανονισμού η βιομηχανία είναι έτοιμη να υποβάλει ε, φακέλους προϊόντων προς έγκριση, όμως πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα σε λειτουργία. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους κοινοποιημένου ε, οργανισμούς. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί θα πρέπει να, έχουν, να αναφέρονται εγκαίρως και για να έχουν την δυνατότητα να διεξάγουν αυτήν την διαδικασία πιστοποίησης μέχρι τα μέσα του 2020. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 58 κοινοποιημένου οργανισμούς ε, που έχουν διαπίστευτεί, όμως μόνο ένας από αυτούς πληρεί τις προποθέσεις για τον νέο κανονισμό. Νομίζω πως φαίνεται πως ε, εδώ θα υπάρξει πρόβλημα. Τα μέτρα για, το, για τη μεταβατική περίοδο, την περίοδο χάριτος ας πούμε, που ε, θα διευκολύνει την ομαλή μετάβαση δεν αρκούν. Δεν συμπεριλαμβάνουν αρκετά προϊόντα της ε, κατηγορίας 1, τα οποία για πρώτη φορά θα χρειάζονται ε, πιστοποίηση από κοινοποιημένο οργανισμό. Μιλάμε για πολλά επαναχρησιμοποιούμενα χειρουργικά εργαλεία. Λίγα παραδείγματα μόνο σας ανέφερα, υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα. Θεωρούμε πως πρέπει να παρασχεθεί λύση άμεσα από τα τρία όργανα, έτσι ώστε η βιομηχανία να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις ε, νέες πιο αυστηρές απαιτήσεις ε, και με τον ε, νέο κανονισμό. Ωστόσο, ίσως δεν, δεν θα περιμένουμε τόσο πολύ μέχρι να δούμε τις συνέπειες όλων αυτών. Ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα αποτελούσε δυνητικό πρόβλημα. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει χιλιάδες ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ευρώπη, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως αρμόδια αρχή από τις 30 Μαρτίου και μετά, εφόσον αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από την αλυσίδα εφοδιασμού, από τα νοσοκομεία, από τους ασθενείς. Η έλλειψη λοιπόν ενός τέτοιου συστήματος ε, ετοιμότητας ε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο χρειάζεται επίλυση αμέσως. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι η βιομηχανία θα συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της στο ακέραιο και με χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ντομακέ, που είναι αναπληρωτής διευθυντής, ε, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής.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 Θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη μία τέτοια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερομένους. Μας προσφέρει και μια ευκαιρία να μεταφέρουμε τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι να διατίθεται στην αγορά ασφαλής, ε, ε, ε, ασφαλή γιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλή και εξυπηρετούν το σκοπό του. Υπάρχουν υψηλέ απαιτήσει όσον αφορά την ασφάλεια αυτών των βοηθήματων. Και παρά τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ε, βοηθήματα από τα πιο ασφαλή σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μία σειρά υποθέσεων, περιπτώσεων, προβλημάτων στο παρελθόν σχετικά με την έγκριση που δείχνουν κάποιες ελλείψεις στο σύστημά μας. Και σκέφτομαι καταρχάς το σκάνδαλο του 2012. Έκτοτε, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εργαστεί σκληρά για να βελτιώσουν την ε, ποιότητα των γιατροτεχνολογικών βοηθημάτων ε, στην αγορά. Χρειαζόμαστε καταρχάς ε, κάποιες άμεσες βελτιώσεις του συστήματος και δεύτερον χρειαζόμαστε μια γενική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και επανεξέταση των νομοθετημάτων που υιοθέτησαν οι συνομοθέτες την άνοιξη του 2017 λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουν γίνει τώρα, Νομίζω ότι το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πιο αυστηρούς τους κανόνες όσον αφορά την κοινοποίηση και τους εθνικούς φορείς για την έγκριση των γιατροτεχνολογικών βοηθημάτων. Έχει αυξηθεί έτσι ο έλεγχος ποιότητας, κάτι που οδήγησε και σε μείωση των ε, φορέων ε, κοινοποίηση από 80 σε 58. Επίσης έχουμε νέες ρυθμίσεις όσον αφορά τις εθνικές αρχές. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε το δρόμο για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και με την έγκρισή του από τους συνομοθέτες θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2020 για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και το 2022 για τα ε, in vitro ε, βοηθήματα. Πιστεύουμε ότι η νέα νομοθεσία θα οδηγήσει σε σημαντικά πλεονεκτήματα. Θα έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τους κοινοποιημένους φορείς. Ε, για παράδειγμα, η αρμοδιότητα και η αμεροληψία θα εφαρμοστούν με πιο αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Επίσης, ε, θα έχουμε πιο αυστηρή εποπτεία στην ε, εσωτερική αγορά. Κλινικές δοκιμές ε, για προϊόντα υψηλού κινδύνου με συμμετοχή μια ομάδας εμπειρογνωμόνων. Έτσι λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες των προϊόντων αυτών. Και Τρίτον, ο νέος κανονισμός θα επιφέρει περισσότερη διαφάνεια. Μέχρι το Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, ε, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα γιατροτεχνολογικά βοηθήματα που ε, τοποθετούνται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά λοιπόν θα έχουμε εκθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Αυτό είναι σημαντικό επίτευγμα, διότι αυτή τη στιγμή τέτοιες πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά από τις εθνικές αρχές. Σημαντικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Euromed, για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με διορθωτικές δράσεις των ε, κατασκευαστών και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιους από τους ισχυρισμούς που ακούστηκαν κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των ερευνών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάποια ΜΜΕ πιστεύουν ότι η βιομηχανία επηρεάζει τις επιλογές πολιτικής μας εις βάρος ε, της υγείας και της ασφάλειας. Στη αναθεώρηση της νομοθεσίας, όπως ε, την, ε, ε, την αντιμετωπίσαμε αυτήν όπως όλες τις άλλες νομοθετικές προτάσεις. Ακούσαμε τα στοιχεία από όλες τις ομάδες που θέλουν να υποβάλουν τις απόψεις τους με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Είτε μιλάμε για τη βιομηχανία, ομάδες ασθενών, πολίτες. Είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε όλες τις απόψεις που εκφράζονται. Και ευχαρίστως τις αξιολογούμε και καταλήγουμε σε διάφορες επιλογές, εκ των οποίων τελικά επιλέγουμε μία ως βάση της πρότασής μας. Αυτή λοιπόν είναι η κανονική νομοθετική διαδικασία και η νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ε, Κατόπιν έχουμε την ε, βάση δεδομένων ε, Euromed. Υπόθηκε ότι δεν είναι αρκετά ανοιχτή και διαφανής όσο θα έπρεπε. Ναι, πράγματι συζητάμε ακόμη το εύρος των πληροφοριών ε, που θα διατίθενται και πιθανότατα να μην δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες, αλλά αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε πολύ, καλές, σε πολύ σωστές αιτίες. θα πρέπει να διαπιστώνεται εάν τα προβλήματα οφείλονται σε κακή λειτουργία του γιατροτεχνολογικού βοηθήματος ή αν οφείλονται σε άλλες αιτίες. Θέλουμε να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών και όχι παραπληνητικές πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη ώστε όλοι να μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες για τα τεχνολογικά βοηθήματα και τη χρήση τους. Θα πρέπει να έχουμε ένα απόλυτα λειτουργικό σύστημα και νομίζω ότι μας ενδιαφέρει κυρίως η ασφάλεια των ασθενών και δεν μας ενδιαφέρει το εμπορικό ε, κέρδος όπως ε, υπενόησαν κάποιοι. Κλείνοντα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη δουλειά που έχει κάνει η διεθνή Κοινοπραξία Δημοσιογράφων Ερευνητών. Οι ανησυχίε σα ευθυγραμμίζονται με τις ανησυχίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νομοθέτη για να έχουμε σωστή αναθεώρηση της νομοθεσίας. Θέλουμε την πιο ε, ασφαλή και καινοτόμα ε, ε, περίθαλψη υγείας ε, και μας ενδιαφέρει πάντα να αντιμετωπίζουμε αδυναμίες του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη και όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Για να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Είναι όμως μια συλλογική προσπάθεια, απαιτείται συνεχής προσπάθεια. Είναι σημαντική η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω όμως ότι έτσι θα πετύχουμε εγκαίρως να παρουσιάσουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Καλό τους συναδέρφους να σχολιάσουν, να θέσουν ερωτήσεις. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω όχι μόνο εξ ονόματός μου, αλλά και εκ μέρους της κυρίας Μαγκίνης, που δεν μπορούσε εδώ να είναι παρούσα σήμερα και ήταν σκιώδης ε, για τα ιατροτεχνικά. Το γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και καθότι έχουμε την ίδια θέση, επιτρέψτε μου να παρέμβω εξ και των δύο. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά του τομέα αυτού που σώζει ζωές, να το θυμίζουμε, και βελτιώνει και τις ε, ζωές πολλών ασθενών. Έχουμε κάποια κρούσματα ε, απάτης και κάποια κρούσματα τεχνικής αποτυχίας ε, και θέσεις σε αγορά επικίνδυνων προϊόντων, αλλά δεν πρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα για το σύνολο του κλάδου αυτού και των προϊόντων και συσκευών αυτών οι αποκαλύψεις αυτές που μας ε, κάνουν τα implant files μας δείχνουν κάποιες νομοθετικές ελλείψεις οι οποίες είναι πραγματικές αλλά οι οποίες είναι ακριβώς αυτές που ήθελε να διορθώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, βελτιώνοντα και τροποποιώντας τη σχετική νομοθεσία. Όμως δεν περιορίζεται ο ρόλος μας εδώ. Έχουμε ενισχύσει τους κανόνες του ελέγχου και πριν και μετά τη θέση σε εμπορία. Έχουμε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης. Δεν θα το επαναλάβω όλα αυτά τα στοιχεία. Και επομένως θα ήθελα ε, να εκφράσω μια απογοήτευση για την γενίκευση των παρατηρήσεων και των εισηγήσεων αυτών. Ε, μπορούμε να υπογραμμίζουμε κάποια προβλήματα, αλλά όχι να ε, μεταδίδουμε ένα αίσθημα γενικευμένου κινδύνου και πανικού για όλο το κοινό. Ακούσαμε το μέγεθος 5,2 εκατομμυρίων ε, περιπτώσεων στις Ηνωμένε Πολιτείε χωρίς να αναφερόμαστε στο γεγονός ότι η τράπεζα δεδομένων αναφέρονται σε, σε επεισόδια συμπεριλαμβανομένων ασθενών που φέρουν ε, εμφύτευμα, χωρίς όμως να ε, οφείλεται το επεισόδιο αναγκαστικά στο εμφύτευμα. Λοιπόν, ε, για την κυρία Μαγκίνες και για μένα την ίδια, το θέμα είναι η σωστή υλοποίηση των διατάξεων του κανονισμού και φοβούμε ότι οι προθεσμίες δεν τηρούνται Υπάρχει ένα θέμα χρονοδιαγράμματος, υπάρχει το θέμα του Brexit, τι θα συμβεί με αυτό το θέμα αν δεν έχουμε συμφωνία, αν έχουμε άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν αυτές οι συσκευές ε, που ε, ε, πιστοποιούνται από οργανισμούς Βρετανι, βρετανικούς, τι θα γίνει με αυτές τις συσκευές, θα είναι ακόμα διαθέσιμες στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις και επ' αυτόν, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Ντιουφάζη, ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ είμαι πολύ λιγότερο αισιόδοξη από τη συνάδελφο. Επί του κανονισμού αυτού, θα ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους για την έρευνα. Έχουμε προβλήματα διαφάνειας, υπευθυνότητας και σημάτων κινδύνου, προειδοποίησης. Για το θέμα της διακυβέρνησης με την κυρία Γοσμπερέν που ήταν προηγουμένως εισηγήτρια είχαμε συζητήσει για έναν ε, κεντρικό οργανισμό να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Έχουμε τον οργανισμό φαρμάκων. Για τις ε, ιατροτεχνικές συσκευέ είναι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Enterprise, το JRC, το Κοινό Κέντρο Ερεύνης. Ποιος είναι ο υπεύθυνο. Υπάρχει χάος. Επίσης, μιλούμε για επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις συσκευές τις πιο επικίνδυνες. Θα έχουμε διαφάνεια για τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων. Θα έχουμε διαφάνεια για τις μελέτες, ε, τις κλινικές που θα έχουν γίνει για να ξέρουμε ε, κατά πόσον επί τη βάση των αξιολογήσεων θα γίνουν, θα ληφθούν συμπεράσματα. Και επίσης για τους κοινοποιημένου οργανισμούς, για τους πιστοποιημένους οργανισμούς, κοιτάω τη μελέτη ε, την έκθεση της Επιτροπής που λέει ότι κοίταξε τους πιστοποιημένους αυτούς φορείς, για έλλειψη ανεξαρτησίας μιλάει, για δομικά προβλήματα διαρθρωτικά, για θέματα διακυβέρνησης, για θέματα πιστοποίησης του προσωπικού, εξειδίκευσης, αριστείας, εμπειρογνωμοσύνης. Δηλαδή, εάν η πλειονότητα των οργανισμών των φορέων αυτών είναι ιδιωτικοί φορείς, όσο περισσότερο θα έχουν σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσα περισσότερα χρήματα θα έχουν. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτοί που θα κάνουν την πιστοποίηση θα είναι ανεξάρτητοι. Μιλάτε για το Udamed. Θαύμα για την τράπεζα δεδομένων. Ποιος θα διαχειριστεί την τράπεζα δεδομένων. Ποιος. Λέτε δεν θέλουμε να δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες γιατί αυτό θα, θα στείλει σήμα κινδύνου στο κοινό. Πανικού. Μα δηλαδή μιλούμε για το 2019 ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις μελέτες, στις ε, επιστημονικές, στις κλινικές. Δεν είμαστε υπαρκώς ενήλικοι για να τα ξέρουμε αυτά. Ποιος νομίζετε ότι είστε, ποιοι νομίζετε ότι είστε μιλούμε για δευτερογενείς επιπτώσεις επί των εμφυτευμάτων. Ποιος θα δώσει σήμα κινδύνου αν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία υπάρξει μια, ένα κρούσμα. Ποιος είναι υπεύθυνο. Άρα θα είναι οι εθνικοί φορείς και οι οργανισμοί. Κοιτώντα την κατάσταση στη Γαλλία, οι εθνικοί φορείς για την επιτήρηση της αγοράς όπως τους ονομάζουμε, περιορίζουν, ορίζουν μάλλον τους επιθεωρητές. Δηλαδή Πώ θα τα μάθουμε τελικώς όλα αυτά. Εγώ ενασυχώ πάρα πολύ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη. Χρειαζόμαστε έναν υπεύθυνο και διαφανή κεντρικό οργανισμό. Δεν τον έχουμε και μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Ε, όχι, δεν πάνε καλά. Οι δημοσιογράφοι μας λένε ότι οι οργανισμοί πιστοποίησης έχουν δώσει σήμα, έχουν δώσει άδεια και δεν έχουν κάνει τον τεχνικό εξοπλισμό για να κάνουν τις δοκιμές. Δηλαδή όλα αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Δεν νομίζω ότι έχετε ε, ε, λάβει υπόψη σας τη σοβαρότητα του, της κατάστασης αυτής και θα έχετε την ευθύνη αύριο όταν θα έχουμε σκάνδαλα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλαμε να υπογραμμίζουμε το, θέμα της διαφάνειας. Εσείς κάνατε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε τις επιχειρήσεις και όχι την ε, δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Ah, it's time of uh, <laughs> the year. Μάλλον είναι η εποχή. Η κυρία Σέρπρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με ανησυχεί αυτό που ακούω. Στις ε, κάτω χώρες υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και στην Ισπανία επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για τα εμφυτεύματα αυτά. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι ασθενείς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιες ε, συσκευές ευθύνονται για ε, θανάτους ασθενών. Νομίζω πως θα ήταν καμιά κάποια πρόοδος αν ε, δημιουργούταν ένα ταμείο το οποίο θα αποζημίωνε τους ασθενείς που θα είχαν άσχημες ε, επιπτώσεις ε, από την κακή λειτουργία ενός τέτοιου προϊόντος. Οι νέες προδιαγραφές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το Μάιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν προβλέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τα περιστατικά σχετικά με αυτά τα προϊόντα. Τι θα γίνει όμως μέχρι την ε, θέση σε ισχύ οι ασθενείς διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους. Τι θα γίνει λοιπόν, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι. Ήδη το έχω ξαναπεί η γερμανική κυβέρνηση έχει νομοθετήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό το οποίο θα βελτιώσει την διαδικασία ελέγχου των ιατροτεχνολογικών αυτών ε, προϊόντων. Ε, βηματοδότες ας πούμε κτλ. Το Υπουργείο Υγείας των Κάτω Χωρών πέρυσι Ε, κατέστησε σαφές ότι οι γιατροί θα πρέπει να δηλώνουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν στους ασθενείς. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει τη δημιουργία κάποιας βάσης δεδομένων. Και αυτό για μένα σημαίνει ότι τον κίνδυνο διατρέχει ο ασθενής. Τώρα, στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο FDA είναι ο υπεύθυνο οργανισμός για οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα τεχνολογικό προϊόν από, μια, από, από ένα αναπηρικό μαξίδιο μέχρι ένα βηματοδότη. Οι Αμερικανοί έχουν βάση δεδομένων, έχουν στοιχεία που πάνε πίσω πάρα πολλά χρόνια και οι ασθενείς οι επιστήμονες, οι γιατροί, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων. Δεν είναι περιορισμένο το κοινό που έχει πρόσβαση σε αυτήν. Άρα δηλαδή, με λίγα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο, όμως ε, αφορά όλους μας και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, ακριβώς διότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Οφείλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους πολίτες, διότι είναι τρομακτικό ε, να σκέφτεται κανείς ε, ποιου κινδύνους ε, διατρέχουν οι ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι εμείς ως νομοθέτες πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους δημοσιογράφους οι οποίοι διενήργησαν αυτήν την έρευνα για τα εφτεύματα, διότι μας δίνει στοιχεία, ενδείξεις για έναν τομέα για τον οποίο δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτό της έλλειψης διαφάνειας, της έλλειψης ιχνηλασιμότητας για την καλή λειτουργία των συσκευών, στοιχεία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, στοιχειοθετούν, συνθέτουν μια εικόνα αρκετά ανησυχητική για την προστασία της δημόσιας υγείας. Εγώ άκουσα παροσεκτικά όλες τις ε, τοποθετήσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι και ο κλάδος ε, κάνει βήματα προς τα εμπρός ώστε να εγγυηθεί την υγεία των πολιτών, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο εμείς. Έχουμε ένα βέβαιο δεδομένο ότι δηλαδή η ασφάλεια μιας συσκευής ιατροτεχνολογικής πιστοποιείται από οργανισμούς ιδιωτικούς και κερδοσκοπικούς, όχι όπως γίνεται δηλαδή με τα φάρμακα, και σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιας τεχνικής συσκευή, αυτά τα κρούσματα δεν συγκεντρώνονται σε ένα μητρό. Δεν υπάρχει λασιμότητα. Αυτά τα χρόνια μάλιστα χάρη και ε, στην πρόοδο της επιστήμης, ε, της τεχνολογίας, ε, έχουμε όλο και περισσότερα κρούσματα δυσλειτουργιών στην Ήπειρό μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ήδη ελέγχθη, η FDA τηρεί δημόσιο αρχείο και δημόσια προσβάσιμο αρχείο. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να είμαστε πίσω σε σχέση με άλλες χώρες. Νομίζω ότι υπό το φως της έρευνας αυτής που διενεργήθηκε θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει οπωσδήποτε μια άμεση τροποποίηση του κανονισμού μέσω της ε, πρόνοιας δημιουργίας εντός της EMA ε, μιας δομής αξιολόγησης των συσκευών αυτών ώστε να υπόκεινται σε πιο άμεση και πληρέστερη παρακολούθηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμεί ω νομοθέτε για να καταλάβουμε ποιε είναι οι αναγκαιότητε προκειμένου να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση για την Γενική Διεύθυνση GROW. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη διαδικασία ορισμού αυτών των κοινοποιημένων οργανισμών. Νομίζω υπάρχει μόνο ένας. Τι μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε να επισπευστεί η διαδικασία. θα καταφέρετε να τηρήσετε τις ε, προθεσμίες για τον ε, ορισμό των κοινοποιημένων οργανισμών και αν όχι τι θα γίνει. Ποιο είναι το σχέδιο Β σε περίπτωση που δεν ανταπεξέλθετε στο χρονοδιάγραμμα. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε περισσότερα από την DigiGrow γι' αυτό. Τη ερώτηση λοιπόν ολοκληρώνει τον κύκλο των ερωτήσεων και τώρα θα δώσω το λόγο και στους τρεις ομιλητές έτσι ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα που ετέθησαν. Θα σας ζητήσω να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά έκαστος έτσι ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής μας. Ο κύριος Μπάουερς θα ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις. Κάποιοι από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στο σκάνδαλο για τα εμφυτεύματα και είπαν ότι αυτό ήταν μια παρέκτηση μιας ε, βιομηχανίας με πολύ καλή φήμη και που έκανε πολλά θετικά πράγματα. Ε, λοιπόν για εξαίρεση και ότι θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε όλη την βιομηχανία για αυτή την υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι Ε, αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων, διότι και μόνο για τα στήθου στήθους ε, είχαμε πάρα πολλές ιστορίες ε, τρομακριτές. Είναι λοιπόν συστημικό πρόβλημα και συνδέεται με την ελαφρά νομοθεσία, το ελαφρύ καθεστώς που έχουμε στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρθηκε ότι η βιομηχανία αυτή κάνει πολλά καλά. Ναι, τα γιατροτεχνολογικά βοηθήματα βοηθάνε και είναι δύσκολο να μιλάει κανείς ως δημοσιογράφος για τον τομέα αυτό της βιομηχανίας χωρίς ε, να, είναι, να γίνεται άδικος, αλλά... Σαφώς το θέμα δεν είναι πώς ωφελούνται οι ε, ασθενείς ε, είναι ο, ο ε, αναγκαίος κίνδυνος και τα μέτρα που αναλαμβάνει η βιομηχανία τη διαχείριση του κινδύνου αυτού, του αναπόφευτου κινδύνου. Και τα μέλη της MedTech ε, Europe είναι επιχειρήσεις. Όχι καλές επιχειρήσεις, απλά επιχειρήσεις είναι. Και επενδύουμε σε αυτές ε, και δεν έχει νόημα να ξεφύγουμε από το γεγονός ότι μάλλον να βγάζουμε συμπέρασμα από το όφελος στους ασθενείς ότι είναι καλές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στόχο έχουν το κέρδος και πρόκειται για ε, μια βιομηχανία που έχει φήμη για την πολύ επιθετική στάση της ε, στην ε, αγορά και ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε σκάνδαλα και στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν προσπαθήσει να βγάλουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα από το πρόγραμμα Medicare. Δεν λέω ότι είναι καλές κακές επιχειρήσεις, είναι όμως εμπορικές επιχειρήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προσοχή όσον αφορά τη ρύθμιση. Δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το εξή. Αρκετοί θεώρησαν ότι οι δημοσιογράφοι λανθασμένα ισχυρίζονται ότι ε, τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να δημοσιεύονται, διότι δεν είχαν επαληθευτεί όλες οι περιπτώσεις ως συνέπεια ε, του γιατροτεχνολογικού βαθύματος. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από τον τομέα αυτών θα αναγνωρίσουν ε, ότι πολλά τέτοια περιστατικά ε, είναι τέτοια που δεν μπορούν να διαπιστωθούν οι αιτίες. Το ότι δεν μπορεί όμως να καθοριστεί από ακριβώς η αιτία δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική πηγή πληροφοριών για τα γιατροτεχνολογικά βοηθήματα και μάλιστα έχουμε πολλά παραδείγματα προϊόντων που ανακλήθηκαν λόγω πολλών τέτοιων αναφερομένων ε, περιστατικών χωρίς να έχει διαπιστωθεί ε, αναφίβολα η αιτία. για τις... για τις ε, συσκευές ε, Φιντέλης η ανάκληση έγινε λόγω του μεγάλου αριθμού των ε, αναφερομένων περιστατικών χωρίς να έχει διαπιστωθεί αδιαφυσβήτητα η αιτία τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρέχονται αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Περνουσκόνη, παρακαλώ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα σχόλια. Εμείς ως κλάδος εξετάζουμε τον κανονισμό αυτό εδώ και καιρό. Και είναι σπάνιο για έναν κλάδιο της βιομηχανίας να μπει σε μια διαδικασία επικαιροποίησης τροχάδιν και καθότι εξελίσσεται το νομοθετικό πλαίσιο κόμμα. Και νομίζω ότι πολλές από τις διατάξεις δεν είναι κατάλληλες πλέον διότι έχει περάσει πολύ καιρός και η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για τις κλινικές δοκιμές χρειαζόμαστε τρόπους ώστε να παρακολουθούμε καλύτερα την απόδοση, την επίδοση αν θέλετε των συσκευών. Ποτέ δεν ήμασταν κατά του στοιχείου αυτού. Εμείς τη χρειαζόμαστε τη διαφάνεια. Γιατί στο τέλος δεν είναι καθόλου καλό για τον κλάδο μας να έχουμε ειδήσει σχετικά με δυσλειτουργίες και σκάνδαλα. Κάποιες περιπτώσεις λοιπόν έχουν γνωστοποιηθεί, έχουν υποβληθεί. Και βλέπει κανείς ότι ασχολείται το σύστημα με τις περιπτώσεις αυτές. Μετά από κάποια δημοσιεύματα είχαμε μαζικές ανακλήσεις. Ίσως ο τρόπος που εξηγήθηκαν ορισμένα πράγματα να μην ήταν ο καλύτερος δυνατός. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση αναγνώριση του κλάδου ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι, πρέπει να είμαστε διαφανείς. Τώρα κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός, μητρό κτλ. Υπάρχει και για μας κάτι σαν EMA οργανισμός και έχει δύο κεφάλια. Την Εθνική Αρχή και την ε, ε Κομισιόν. Μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο, περίπλοκα, αλλά εν πάση έχουμε δομές. Έχουμε δομές σήμερα που μπορούν και πρέπει να διέπουν αυτά τα πράγματα και μπορούμε και πρέπει να τα βελτιώσουμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έχουμε μια πρόταση σήμερα για νέο κανονισμό και αυτό θα πρέπει να κινηθεί να είναι έτοιμος από τον Μάιο του 20. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία και δεν πρέπει να φοβούμαστε να πούμε ότι από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα που να μπορεί να παρακολουθεί κατά πόσον οι προσδοκίες μας έχουν καλυφθεί και από τον ιατρο, ιατρικό κλάδο και από όλους τους επαγγελματίες που ενέχονται. Αν τα πράγματα δεν κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Άρα χρειαζόμαστε παρακολούθηση. Και μην λέμε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε όλα τώρα. Αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή, να επανέλθουμε σε, σε χρόνια συζητήσεων προτού να κινηθούμε. Προτού εφαρμόσουμε τον νέο κανονισμό. Τον χρειαζόμαστε τον νέο κανονισμό. Για την προστασία των ασθενών και της δημόσιας υγείας και της ασφάλειάς τους. Πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί ο κανονισμός και να δρούμε με διαφάνεια. Και να συζητήσουμε και για την UDAMED, την τράπεζα δεδομένων. Δεν φοβόμαστε την διαφάνεια και δεν πρέπει να την φοβόμαστε. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε εμείς. Μην το σκέπτεστε. Είναι αδύνατον ούτως ή άλλως στον σημερινό κόσμο να κρύψει κανείς τη διαπράγματα λέει ο μιλητής. Αλλά ας τα κινήσουμε αυτό. Γιατί αλλιώς θα είναι απλώς ωραία λόγια. Very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα πάρει το λόγο. Χρειάζεται να εφαρμοστεί νομοθεσία. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσω απαντώντας την ερώτηση σχετικά με το που βρισκόμαστε ως προς την εφαρμογή ε, των διατάξεων για τον ορισμό των κοινοποιημένων οργανισμών. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 45 αιτήσει ε, για ορισμό κοινοποιημένων οργανισμών, 25 ε, αξιολογήσεις διεξάγονται αυτή τη στιγμή από κοινού και θα ξεκινήσουν οι υπόλοιπες πολύ σύντομα. Με βάση αυτά νομίζω πως οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που ε, έχουν καταθέσει αιτήσει, το έχουν κάνει έτσι όπως πρέπει και νομίζω πως τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για όσους κοινοποιημένους οργανισμούς έχουν καταθέσει αιτήσει. Εργαζόμαστε σκληρά λοιπόν και ελπίζουμε όμως να κάνουν το ίδιο και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί στα κράτη-μέλη. Διότι είναι κοινή μα ευθύνη. Η κυρία Γκροστέτ νομίζω ρώτησε ε, κάτι σχετικά με το Brexit. Τι θα γίνει. Βέβαια, δεν ξέρω τι έχει ψηφίσει η Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα και δεν μπορώ να ξέρω πώς θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι ε, όλα τα κράτη-μέλη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και έχουμε δώσει έμφαση στους ε, κοινοποιημένους οργανισμούς ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο και πώς μπορούν να αντικατασταθούν από κοινοποιημένους οργανισμούς στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη. Εξετάζουμε τους ε, κινδύνους ε, πιθανών ελήψεων, εφόσον αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα συγκεκριμένα, συγκεκριμένη κίνδυνοι. Εάν όμως είχαμε εντοπίσει κάποιους κινδύνους, ε, να είστε σίγουροι πως θα είχαμε ξεκινήσει ήδη ε, να δουλεύουμε κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ή σχέδιο Β. Τώρα, ποιο είναι υπεύθυνο, μα ρωτήσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πω ε, καταρχά πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα θεσμό. Υπάρχει το Κέντρο Κοινών Ερευνών. Όμως γενικότερα για την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ είναι κάθε αρμόδια και συνεισφέρει πάρα πολύ στις ε, προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή για να τεθεί σε ο κανονισμός. Τώρα, φυσικά μιλήσατε για διαφάνεια, για εχνηλασιμότητα. Θα ήθελα να σας απαντήσω πως είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή η UDAMED, η βάση δεδομένων, καλύπτει τις ελλείψεις, τα κενά που υπήρχαν. Και νομίζω πως μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις που υπάρχουν ε, και σχετικά με την ε, καταχώρηση των ιατροτεχνικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αλλά και ως προς την... Ε, τον έλεγχο της αγοράς. η πρόσβαση στην πληροφορία και σε αυτή την βάση δεδομένων είναι κάτι που ε, θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές ήταν οι ερωτήσεις που έγιναν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε για να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα Παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και περιμένουμε από τη βιομηχανία να κρατήσει το λόγο της για περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού. Διότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους κύριους δημοσιογράφους και όλους τους ε, συναδέλφους. Και εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Περνάμε τώρα στην πρόταση για πράξη της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την ενίσχυση της συλλογής πλάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία πρόταση από τις 18 Δεκεμβρίου από τον κύριο Καπούτο, την κυρία Πίρικ και άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Η Επιτροπή μας είναι η καθήλυνα αρμόδια. Έγινε γνωστό αυτό στις 16 Ιανουαρίου. Σήμερα λοιπόν εξετάζουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη έτσι ώστε να επιτρέψουμε στους συντάκτες της πρότασης να την παρουσιάσουν ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων. προβλέπετε να ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό εντός τριών μηνών μετά την αναπομπή στην Επιτροπή. Αφού αποκτήσουν τη δυνατότητα οι συντάκτες να παρουσιάσουν την πρόταση στην Επιτροπή. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στον κύριο Καπούτο για περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών ε, που συνδέονται με επεισόδια παθολογίας ε, σχετικών με το πλάσμα του αίματος. Είναι αυξημένη η ανησυχία η σχετική και επομένως τα φαρμακευτικά σκευάσματα θα πρέπει να λειτουργούν, ε, καλούνται μάλλον να λειτουργήσουν με, με μια πρώτη ύλη όλο και πιο δύσκολα ευρέσιμη σε άριστη ποιότητα. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πλάσματος αίματος εισάγεται από την Αμερικανική αγορά όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ε, αγορά η οποία διέπεται, ρυθμίζεται από την FDA και επομένως εξαρτώμεθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από παράγοντες που διαφεύγουν του ελέγχου μας. Η Κομισιόν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη διαθεσιμότητα παραγωγής πλάσματος για τα σκευάσματα που απαιτείται εκεί όπου έχουμε διαγνώσεις παθολογιών όπως η ομοφιλία, ε, ε, συγκεκριμένες νόσους και σύνδρομα αυτοάνοσα και γι' αυτό προτείνουμε αυτό το Union Act και μια αναθεώρηση ε, της οδηγίας για το αίμα και γενικώ το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να διέπεται όλη η, το σύνολο του όγκου της δωρεάς αίματος σε όλα τα κράτη-μέλη. Εύχομαι πραγματικά, Πρόεδρε, ότι στην επόμενη συνάντηση συντονιστών θα, μπορούσαμε, θα μπορέσουμε να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή που αποσκοπεί ε, στη διαφύλεξη της προστασίας υγείας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο ως συντάκτη, συντάκτρια μάλλον, κυρία Σάιν Πέρικ. Πρόεδρε. Είναι πολύ θετική η πρόταση αυτή. Το πλάσμα χρησιμοποιείται σε πολλές θεραπευτικές αγωγές και ασθενείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ασθένειες που χρειάζονται τέτοιες θεραπείες. Το 40% του πλάσματος που χρειάζεται εισάγεται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχουμε καθόλου έλεγχο τις ε, τροφοδοσίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, πληρώνονται ε, οι δωρεές πλάσματος, αλλά όταν κάποιος το κάνει αυτό για τα χρήματα, μπορεί να μην είναι ειλικρινής όσον αφορά την υγεία τους. Ελέγχεται βέβαια το πλάσμα, κάποιες ασθένειες όμως δεν μπορούν να εντοπιστούν τόσο νωρίς. Το πλάσμα που καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Στην αγορά των κάτω χωρών χρησιμοποιείται στο βαθμό που είναι δυνατόν πλάσμα από ε, Ολλανδούς, αλλά δεν έχουμε αρκετό. Έτσι κάποιο τμήμα του πλάσματος που χρησιμοποιείται προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καλύτερο λοιπόν ε, να γίνεται καλύτερη συλλογή πλάσματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για λόγους ανοσολογίας ε, συλλέγεται το πλάσμα και η ζήτησή του αυξάνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει ομάδα εργασίας εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζει την χρήση του πλάσματος ως πρώτη ύλη. Αυτό όμως δεν αρκεί. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το θέμα αυτό. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ασφαλής μέθοδος ε, συλλογής του πλάσματος ε, είναι δωρεάν. Είναι δύσκολο όμως να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό ε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις ώστε να έχουμε αρκετό πλάσμα χωρίς ε, να ε, πληρώνουμε τους δωρητές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην εξαρτώμαστε από το πλάσμα από τις ΗΠΑ και γι' αυτό θα ήθελα να στηρίξω αυτή την πρόταση. Κύριε Κροστέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με πολλές από τις παρατηρήσεις των συντακτών ε, γνωρίζω καλά το θέμα των προϊόντων αίματος. Ε, πρόκειται για ε, μια πράξη που είναι απολύτως απαραίτητη και πολύτιμη, αλληλεγγύης για τους πολίτες μας, αλλά το, η πρώτη προτεραιότητα του συστήματος συλλογής θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των, του μεγαλύτερου αριθμού των δωρητών, είτε των δεκτών του πλάσματος. Όμως, όπως λέγει η μελέτη, έχουμε ένα πρόβλημα διαθεσιμότητος. Γιατί έχουμε μια φιλοδοξία ανεξαρτησίας σε προϊόντα αίματος και πλάσματος, γιατί προς το παρόν είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από το αμερικανικό προϊόν, το αμερικανικό πλάσμα και εκεί υπάρχει μια στρατηγική εξάρτηση. Ήθελα λοιπόν να επιμείνω στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε την δική μας κατεύθυνση, το δικό μας άξονα επί τη βάση αρχών ανθρωπιστικών και αλληλεγγύης με τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που θα πρέπει να είναι να διέπει απολύτως την συλλογή του πλάσματος που γίνεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ψευδός σωστή και δίκαιη ιδέα η αμοιβή που θα πρέπει να δίδεται στους δωρητές, οδηγεί σε αντιπαραγωγικές ε, ε, τάσεις ε, και συμφωνώ απολύτως και προσυπογράφω τους, ε, την μελέτη και τους δύο συντάκτες το συμπέρασμα αυτό. Θα ήθελα όμως να επιμείνω και ως προς την αναγκαιότητα για την Ευρώπη να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία εδώ. Μιλούμε για στρατηγική αυτονομία για την προστασία στα θέματα αμήνης και ασφάλειας εάν κάποια μέρα συμβεί κάτι σημαντικό, μεγάλης κλίμακος στην Ευρώπη ή στον κόσμο, εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε μας πούνε δεν σας εξάγουμε άλλο, το χρειαζόμαστε εμείς το δικό μας, τι θα κάνουμε στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μικρής κλίμακος οργανωμένη διαρθρωμένη συλλογή στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το σκεπτούμε αυτό. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να οργανώσουν καλύτερα την συλλογή του πλάσματος πώς θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα να αξιοποιήσουμε την, ε, τους, ε, την, την κίνηση των δωρητών, την προσφορά τους. Όπως είπε και η συνάδελφος. Επομένως πραγματικά ε, πρέπει να κοινοτομήσουμε εδώ. Θα πρέπει να κοινοτομήσουμε προκειμένου να, πάμε, να υπερβούμε το παρόν πλαίσιο. Όμως θα ήμουν πολύ πιο προσεκτική από τους συντάκτες σχετικά με την αναγκαιότητα της αναθεώρησης της οδηγίας για το αίμα. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να βελτιωθούν, αλλά μια νομοθετική επανεξέταση επιφέρει πάντοτε ε, έλλειψη ασφάλειας δικαίου ε, και αβέβαιες κατευθύνσεις. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερπροδραστικοί εδώ, θα πρέπει να διατηρήσουμε κατά νου τα υπέρ και τα κατά, να αναλύσουμε προσεκτικά τον αντίκτυπο του νομοθετικού υφισταμένου πλαισίου, προτού καλέσουμε για αναθεώρηση των πάντων. Ε, και υπό την έννοια αυτή, τα όσα θα μπορούσε να μας πει η Κομισιόν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σέικελ, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, να ευχαριστήσουμε καταρχά ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία που διοργάνωσε. Να πούμε ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει πω οι ασθενεί εξαρτώνται απόλυτα από πλάσμα που εισάγεται από τρίτε χώρε, ιδιαίτερα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αναφέρθηκε ένα ποσοστό τη τάξη του 40%. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα ε, αναφέρουν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το 40% πάρα πολλοί ασθενείς εξαρτούνται από προϊόντα που παράγονται από πλάσμα και σε περίπτωση διακοπής ε, της, ε, του εφοδιασμού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, για τους ασθενείς. Για παράδειγμα, το ξέσπασμα μιας επιδημίας στις ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πλάσμα. Ο ιός Ζήκα, για παράδειγμα, είναι μια πρόσφατη περίπτωση περιστατικού που απείλησε την, ε, την αλυσίδα αίματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ε, δημόσιας διαβούλευσης ε, αναφέρθηκε το θέμα αυτό και το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιες αρχές και από τις δύο πλευρές από την ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησαν να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για το πλάσμα έτσι ώστε να υπάρχουν ε, αυξημένα επίπεδα προστασία, αλλά και για να προστατεύονται οι δωρητέ πλάσματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρακτικά τη συνεδρίασης έχουν δημοσιευθεί, είναι διαθέσιμα και αυτή τη στιγμή καταρτίζεται η τελική έκθεση για την αξιολόγηση αυτή τη άσκηση, έτσι ώστε να δούμε πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις και τι ανησυχίε που έχει γύρει η αξιολόγηση αυτή. Φυσικά θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, παράλληλα, Συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης ε, σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εκείνους για να δημιουργηθεί ένα σχέδιο που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και ε, ως προς τη συλλογή πλάσματος και ένα, ως προς ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που υπάρξουν ελλείψεις ή διακοπή στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ελπίζουμε λοιπόν πολύ σύντομα να έχουμε αποτελέσματα και από τις ε, δύο αυτές ε, δράσεις. Είναι λοιπόν ήδη στο πρόγραμμά μας, ε, γι' αυτό λοιπόν θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρωτού ολοκληρώσω τη σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια ένσταση σχετικά με τις ε, συστάσεις των συντονιστών ε, της 27 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε πως στάσεις έχουν εγκριθεί. Στις 14 Μαρτίου, στις 9 το πρωί στο Στρασβούργο, θα λάβει χώρα επόμενη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.